Right, good afternoon everybody. Καλό απόγευμα σε όλους. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας γιατί θέλουμε να έχουμε χρόνο για ερωταπαντήσεις. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Επίτροπο Αλμούνια Η τελευταία μας συνάντηση με τον Επίτροπο έγινε στις 5 Οκτωβρίου στη δημόσια κρόση για τις κρατικές ενισχύσεις και στις και το 2011 θα επαναλάβουμε το εγχείρημα αυτό. Αλλά σήμερα είναι μαζί μας για να μα κάνει κομισιόν του χρόνου που θα Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ που με ξανακαλέσατε στην Επιτροπή αυτή Οικονομικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να σας πω πράγματι πως βλέπω να διαμορφώνται οι εργασίες στον τομέα του ανταγωνισμού για το 2011. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, θα υιοθετήσετε το ψήφισμα για την ετήσια έκθεσή μας το 2009. Γι' αυτό ξεκινώ λέγοντας ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα και ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμβολή σας, πολλών από εσά και ιδιαίτερα του κυρίου Έπινγκ που ήταν εισηγητής. Ας πω λοιπόν τώρα μερικά πράγματα για το πρόγραμμα εργασιών του 2011. Αρχίζουμε με τα καρτέλα. Ο αγώνας μας ενάντια στα καρτέλ είναι κεντρικός της εργασίας μας, ιδιαίτερα αυτούς τους δύσκολους καιρούς που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ζημιώνεται περισσότερα ή περισσότερο η οικονομία μας λόγω των πρακτικών των καρτέλ. Πήραμε έξι αποφάσεις φέτο για εναντίον καρτέλ ε, ενάντια σε 12 μίζονες αεροπορικές εταιρείες και επιβάλαμε πρόστιμα σχεδόν 800 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά τα μεγάλα πρόστιμα Βέβαια θα προτείνουμε και άλλες αποφάσεις σχετικά με καρτέλ πριν από το τέλος της χρονιάς και το 2011. Τα μεγάλα πρόστιμα πάντως της τελευταίας μας ε, απόφασης οφείλονται στην εξή λογιστική. Θέλουμε ψηλά πρόστιμα για να αποτρέψουμε να αποτρέπουμε συμπεριφορές ε, του ανταγωνισμού αλλά να μην είναι τόσο ψηλά τα πρόστιμα και όλο τους ώστε να αναγκάζονται επιχειρήσεις να κλείνουν. Η γραμμή βέβαια μεταξύ το, το να ακολουθήσουμε αυτά τα κριτήρια, η γραμμή μεταξύ το μεν και το δε δεν είναι εύκολο να χαραχθεί υπό τις παρούσες συνθήκες, αλλά ε, η Κομισιόν συνεχίζει να αγωνίζεται και να επιβάλλει μέτρα ούτως ώστε να μην... Ε, ε, συνεχίζονται παράνομες πρακτικές. Τώρα έρχομαι στον τομέα του αντιτράστ. Ε, ή θέλουμε επιχειρήσεις που παράγουν τα καλύτερα προϊόντα και τις καλύτερες υπηρεσίε στις καλύτερες τιμές. Και όταν και η ενέργεια, δράση που αναλαμβάνουμε σχετίζεται με πολύ σημαντικούς κλάδους όπως τεχνολογία, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, συστήματα πληρωμών κτλ. Ιδιαίτερα στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και τεχνολογίας τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και τα, η είδηση που σας παρουσιάζω σήμερα είναι ότι ξεκινήσαμε την επίσημη διαδικασία για έρευνα σχετικά με το Google. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, θέλω να μην παρεξηγηθώ, είναι πολύ νωρί. Εκείνο που κάνουμε όμως είναι να ερευνήσουμε σε βάθος κάποιες ανησυχίες που υπάρχουν. Στον τομέα της ενέργειας ε, έκλεισε η έρευνα που κάναμε το 2007. Είδαμε ότι υπάρχουν προβλήματα ε, και πρέπει ε, να δώσουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε κάποιες ενέργειες πια για να δώσουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε τις εθνικές αγορές του ανταγωνιστές και να επιτρέψουμε στους καταναλωτές να έχουν ε, εναλλακτικές λύσεις. Εκδώσαμε δύο αποφάσεις σχετικά με διορθώσεις που πρέπει να γίνουν και από εκεί και πέρα ε, το ίδιο πράγμα κάνουμε και για την απελευθέρωση των αγορών τηλεπικοινωνιών. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις για την Πολωνία και τη Σλοβακία. Επίσης προσπαθούμε να αναλάβουμε δράση και στον τομέα των συστημάτων πληρωμής. Μετά από τη συμφωνία με τη Mastercard το 2007 ε, ελέγξαμε την Visa Europe και συνεχίζουμε να ερευνούμε την περίπτωση. Ε, Επίσης ξεκινήσαμε δουλειά σχετικά με τους, μαζί με τον Επίτροπο Μπαρνιέ για να ε, διασφαλίσουμε ότι η ενιαία Ευρωπαϊκή Περιοχή Πληρωμών είναι πλήρης και προωθεί τον δίκαιο ανταγωνισμό, τον Χριστό ανταγωνισμό. Τώρα, πέρα από τα θέματα αυτά των καρτέλ και των υποθέσεων αντιτράστ προσπαθούμε να δούμε εάν ε, υπάρχουν δυνατότητες ε, να βελτιώσουμε και τις διαδικασίες που ακολουθούμε κατά τις υποθέσεις αυτές και ελπίζουμε του χρόνου να προτείνουμε τις βέλτιστες πρακτικές και τις διαδικασίες αντιτράστ. Προχωρούμε στις συγχωνεύσεις. Ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει οι επιχειρήσεις της να είναι παγκόσμιοι πρωτοπόροι παγκοσμίω. Αλλά για να γίνουν πρωτοπόροι παγκοσμίω θα πρέπει να γίνουν πρώτοι στην Ευρώπη πρώτα, στην ευρωπαϊκή αγορά. Και βεβαίω ε, αυτό επηρεάζει τις συγχωνεύσεις η ύφεση την οποία ζήσαμε, ζούμε ε, βλέπουμε ότι επηρεάζει τις συγχωνεύσεις το 2010 παραδείγματος χάρη είχαμε ε, μελετούμε μοναχά 260 κοινοποιήσεις όπως και το 2009 που πράγμα που είναι δύο τρίτα μόνο από τις κοινοποιήσεις του 2007. Το 2010 είχαμε μόνο τέσσερις έρευνες δεύτερης φάσης, ε, Unilever Sara Lee και Syngenta Monsanto που έκλεισαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ η υπόθεση Ολυμπιακής Aegean θα κλείσει τον Ιανουάριο. Όσο προχωρεί η οικονομική ανάκαμψη, τόσο θα αυξάνεται και πάλι ο αριθμός των κοινοποιήσεων για συγχωνεύσεις. Τώρα για τις κρατικές ενισχύσεις. ξέρουμε ότι μάλλον αύριο θα υποβάλω στο Σώμα των Επιτρόπων ε, το, ένα βαθμολόγιο για τις κρατικές ενισχύσεις και θα δείτε ότι ε, οφείλονται οι περισσότερε περισσότερες κρατικές ενισχύσεις στην υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ε, για τους άλλους τομείς τα πράγματα είναι μάλλον σταθερά αντίκτυπος και επιπτώσεις. Το ψήφισμά σας για την, για την ετήσια έκθεση για τον ανταγωνισμό ζητεί από την Κομισιόν να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους αντικτύπους αυτών των μέτρων είναι γεγονός ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση αυτή αλλά κυρίως την ευθύνη την έχουν οι εθνικές αρχές για την εφαρμογή αυτών των μέτρων δεν Εμεί θα σα παρουσιάσω, ζήτησα από τι υπηρεσίε μου να ετοιμάσουν μία μελέτη για το, το 2011, αλλά βεβαίω δεν μπορούμε να μπούμε στι λεπτομέρειε, τι λεπτομέρειες που ενδεχομένω να θέλετε να δείτε. Τώρα, για το εξαιρετικό καθεστώς το, των κρατικών α, ενισχύσεων που ξεκίνησε όταν ξεκίνησε και η κρίση βεβαίως μιλάμε για εξαιρετικό καθεστώς που σημαίνει εξορισμό ότι δεν θα συνεχιστεί ε, δεν θα διανυστεί στο μέλλον τώρα όμως έφτασε η στιγμή να προετοιμάσουμε μια βαθμιαία επιστροφή κανονικές συνθήκες λειτουργίας αγοράς, διβαθμιές συνθήκες γιατί φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάκαμψη αλλά υπάρχει και μια κάποια αβεβαιότητα για το κατά πόσον θα συνεχιστεί αυτό. Αύριο θα προτείνω στο Σώμα των Επιτρόπων την ε, παράταση κάποιων από τα προσωρινά μέτρα που πήραμε το 2011 γιατί χρειάζεται αλλά από εκεί και πέρα θα καταργηθούν βαθμιαία τα μη αναγκαία και απαραίτητα μέτρα θα συνεχίσουμε όμως να, προσπαθήσουμε, να προσπαθούμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας και τις τράπεζές μας πιστεύουμε ότι αν τα πράγματα πάνε καλά θα επανέλθουμε στο κανονικό καθεστώς για τις κρατικές ενισχύσεις από την 1η του Γενάρη του 2012. Και για αυτή την επιστροφή στις κανονικές συνθήκες με μεγάλη χαρά θα συζητήσω μαζί σας αργότερα. Τώρα, τι άλλο όχι θα κάνουμε το 2011. Θα αναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες. Παραδείγματο χάρη την ποσοτική έκφραση των ζημιών λόγω συμπεριφοράς αντιτράστ, κάποια δράση στον τομέα της, ε, των εκπομπών, ε, αναθεώρηση του καθ το κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, στη, στα ναυπηγεία, στις κρατικές ενισχύσεις για τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες. Και να σας δώσω τρία παραδείγματα για το τι θα κάνουμε το 2011. Πρώτα πρώτα, αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Είναι η πρώτη περίπτωση, οριζόντια οι κανόνες ε, συνεργασίας, το δεύτερο παράδειγμα και μετά η συλλογική προσφυγή είναι το τρίτο παράδειγμα. Λοιπόν, για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος κομισιών το 2005 ε, ε, μια δέσμη μέτρων για να υπάρχει μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα για τις ε, υπηρεσίες αυτές. Το 2011 θα αναθεωρήσουμε τη δέσμη αυτή μέτρων για να κάνουμε διορθώσεις. Η αναθεώρηση θα βασίζεται στις εκθέσεις που έκαναν τα κράτη-μέλη και στα αποτελέσματα της δημόσιας διαβουλευση που έκλεισε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Θα ήθελα να ξεκαθαριστεί ακριβώ ιδιαίτερα η διαφορά μεταξύ υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντο. και πότε επιτρέπεται η χρηματοδότηση ε, που γίνεται πότε η χρηματοδότηση από το δημόσιο τομέα ε, θεωρείται κρατική ενίσχυση. Θα πριν να ελπίζουμε ότι και το Σώμα των Επιτρόπων θα εγκρίνει σχετικές αποφάσεις αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας ενημερώσουμε στις ε, αρχές επόμενης χρονιάς. Τώρα για τους οριζόντιους κανόνες συνεργασίας θέλουμε η και δύο πράγματα ο ορισμός προτύπων standards και η ανταλλαγή πληροφοριών να είναι βασικά σημεία αυτών των κανόνων ε, που θα εγκρίνουμε του χρόνου ελπίζουμε τις κατευθυντήριες γραμμές να τις εγκρίνουμε πριν από το τέλος της χρονιάς και δύο λόγια ακόμη για αυτό που ονομάζουμε private enforcement μαζί με τους συναδέλφους Ρέντινγκ ε, και Νταλή ε, υποβάλαμε μια, ένα ενημερωτικό σημείο μας στους υπόλοιπους επιτρόπους σχετικά με πρωτοβουλίες που προτιθέμεθα να αναλάβουμε για να βοηθήσουμε συλλογικές προσφυγές ούτως ώστε να μην έχουμε κατάχρηση της προσφυγής στο μηχανισμό διευθέτησης διαφορών. Σαν πρώτο βήμα θα ξεκινήσουμε μια δημόσια διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους και αν τα πράγματα πάνε καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, αποφασίσει μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση το 2011 και θα υποβάλω και συγκεκριμένη πρόταση μέσα σε αυτό το πλαίσιο για την διόρθωση των ζημιών αποζημίωση λόγω συμπεριφοράς αντιτράστ. Σας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει πλήρως και θα ενημερώνεται στα χρονικά διαστήματα για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very much, um, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα σας διαβάσω τα ονόματα των εγγεγραμμένων που επιθυμούν να θέσουν ερωτήσεις και θα προτείνω πάλι να απαντάω Επίτροπο σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά. Μία ερώτηση, μία απάντηση. Έχω λοιπόν στον κατάλογο. Jose Garcia Magallo, uh, Andreas Schwab, uh, Ramon Tremosa, Sophie Infelt, Werner Langen, Philippe Lamberts, Vicky Ford, Antolin Sanchez, Prozedo. Anybody else want to come in? Wave now. Okay, so Jose. Ο Ζωζέπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πάντα έχουμε ταχθεί υπέρ του fair play με τον επίτροπο, το συγκεκριμένο επίτροπο. Γιατί είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής και είναι υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο του ανταγωνισμού. Στις 26 Νοεμβρίου κάνατε ορισμένες δηλώσεις όπου που αναφέρατε ότι η Ισπανία δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει αυτά ε, στα οποία, τα οποία είχε υποσχεθεί. Την επόμενη ημέρα ο πρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι θα έπρεπε εσείς να επικυρώσετε τις δηλώσεις σας. Σήμερα έχουμε τη δήλωση της Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, γιατί δεν πρέπει να ξέρουμε ότι τα spreads μας φτάσανε τα 300, τις 300 μονάδες μετά από τις δηλώσεις Μέρκελ ότι οι ιδιωτικοί επενδυτές θα πρέπει να συμμετάσχουν στα σχέδια διάσωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αποδυναμώνεται και η κατάσταση και το ευρώ το ίδιο. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο βλέπετε ένα συσχετισμό όλων αυτών για να μην καταλήξουμε σαν το Τιτανικό. Ελπίζω να απαντήσετε με την ακρίβεια και την γενεοδορία που σας ε, χαρακτηρίζει. Επικυρώνεται ότι υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα της Ισπανίας να εφαρμόσει τα σχέδια, τα προγράμματα που είχε ορίσει. Υπάρχει σχέδιο Β. Και ε, ε, αν λάβουμε υπόψη και τους ε, κερδοσκόπους που επιτίθενται κατά του ευρώ, θεωρείται ότι από το 2013, όπως είπε η Καγκελάριος, εφόσον θα συμμετάσχουν και οι ιδιωτικοί επενδυτές στο σχέδιο διάσωσης, υπάρχει λύση απάντηση. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον και προσοχή την εξέλιξη των αγορών τις τελευταίες ημέρες. Θα πρέπει να είμαστε συνετοί ως προς τη δημόσια αντίδρασή μας για την κατάσταση της αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν όλοι, και υπογραμμίζω όλοι, να είμαστε σαφείς, να είμαστε συντονισμένοι ως προς τα μηνύματα που αποστέλουμε και τις δημόσιες απόψεις μας, έτσι ώστε αποφασιστικά να δράσουμε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αποφάσισαν όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, ως προς την Ισπανική κυβέρνηση, όπως είπα στις δηλώσεις μου και επαναλαμβάνω σήμερα, η Ισπανική κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει, δηλαδή προχωρά στην φορολογική ενοποίηση και το χρηματοοικονομικό σύστημα ως προς τις τράπεζες αποταμιεύσεων και όπως τόνισε το Σάββατο και ο πρόεδρος της κυβέρνησης, θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το συνταξιοδοτικό σύστημα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το δημόσιο χρέος πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Άρα η Ισπανική κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά το κάνει με αποφασιστικότητα. Και νομίζω γι' αυτό ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την Ισπανία. Eh, Πιστεύω ότι στο τέλος της εβδομάδας θα υπάρξει υποστήριξη και από το Συμβούλιο και η Ισπανία καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να υπερασπιστούμε το ευρώ έναντι επιθέσεων της αγοράς και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε κατά ευφύ τρόπο όπως είπε το ΕΚΟΦΗΝ, η Ευρωομάδα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό αφορά και τη θέση της ΕΚΤ έτσι ώστε να βελτιώσουμε την λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως ισχύει στην περίπτωση της Ελλάδας, της Ιρλανδίας τώρα τελευταία, για να μπορέσουμε να ορίσουμε προτεραιότητες, νέες προτεραιότητες για την ΟΝΕ. Αυτό αφορά και τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που ήταν εκτός ελέγχου πριν από την κρίση. Το Κοινοβούλιο τάσεται, από όσο γνωρίζω, υπέρ της οικονομικής ρύθμισης μέσα στα πλαίσια ενός γενικότερου συντονισμού και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους κλειδονισμούς της αγοράς κατά αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σβάμπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας συγχαίρω κύριε Επίτροπε για το γεγονός ότι ξεκινήσατε επισήμως την διαδικασία καρτέλ κατά του Google. Κάτι που έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο εδώ και καιρό. Δεν πρόκειται για κάποια πρώιμη καταδίκη, αλλά αναγνώριση των υποθέσεων ότι ενδεχομένω η κωδικοποίηση της μηχανής έρευνας του Google δεν λαμβάνει υπόψη ορισμένα στοιχεία που θα έπρεπε να λάβει. Και αναμένω βεβαίως εγώ με μεγάλο ενδιαφέρον την διευκρίνηση του θέματος. και την έρευνα που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω το χρωστάμε στους πολίτες μας να ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό, διότι δεν κατανοούν ποιες λειτουργίες του Google κρύβονται πίσω από αυτή τη μηχανή έρευνας. Λοιπόν, αυτό θα το δούμε. Αυτά που ήδη είδαμε και χαίρομαι για τα όσα είπατε για τα καρτέλ ε, στην, ε, στο θέμα 2 της ομιλίας σας, ότι δηλαδή η, ε, τα πρόστιμα πρέπει να είναι πολύ υψηλά για να έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα, χωρίς ταυτόχρονα να είναι τόσο ψηλά, ώστε να οδηγούν σε οικονομικές δυσχέρειες της επιχείρησης. Νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα. Νομίζω επίσης ότι την πολιτική αυτή πάντοτε την ε, ε, υπεστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ρωτώ, γιατί βρίσκει τόσο δύσκολο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σφυριλατήσει τα νομικά κείμενα που θα περιλαμβάνουν αυτήν την αρχή την οποία βρίσκουμε και εσείς και εμείς σωστή και στις guidelines, ακόμα καλύτερα και στον κανονισμό για το ε, θέμα. Και νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερη ερώτηση και τελευταία. Μιλήσατε για την πράσινη βίβλο ή για τη νέα διαβούλευση για τις συλλογικές αγωγές αποζημιώσεων. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατήθηκε από το αρχικό σχέδιο και αναζητεί τώρα νέα λύση που θα επιτρέψει αφενός να κάνουν συλλογικές δράσεις οι καταναλωτές, ταυτόχρονα όμως κάνει κάθε προσπάθεια αποφυγής του να έρθουν εδώ και να καθιερωθούν αμερικάνικα πρότυπα ή σχέσεις. Thank you Ο Επίτροπος, ευχαριστώ κύριε Σφάμπ. Οι διαδικασίες που ανοίξαμε επισήμω σήμερα κατά του Google είναι αντιτράστ και όχι καρτέλ, όχι αντικαρτέλ. Αντιτράστ. Είναι σημαντική διάκριση ωστόσο. Ως θα θυμάται η Επιτροπή σας, στις αρχές του έτους λάβαμε τρεις καταγγελίες που εν μέρη αναφέρονταν στη λειτουργία της μηχανής έρευνας και εν μέρη αναφέρονταν στη λειτουργία του διαφημιστικού συστήματος του Google. Αναλύσαμε τις καταγγελίες αυτές σε στενή επαφή με την Google η οποία συνεργάστηκε μαζί μας, μας πρόσφερε πλήθος πληροφοριών τις οποίες εμείς αναλύσαμε. Εν τέλει καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι με τις πληροφορίες που είχαμε στη διάθεσή μας δεν είμαστε εις θέση να απορρίψουμε τις καταγγελίες. Άρα χρειάζεται να διευρύνουμε και να βαθύνουμε την έρευνά μας και νομίζω ότι θα είναι καλύτερα για όλους να γίνει επίσημη η διαδικασία, να ανοίξει επίσημα η διαδικασία δηλαδή και να μην συνεχιστεί σε ανεπίσημη βάση. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο από την αντίδραση του Google στην, στο άνοιγμα της επίσημης διαδικασίας, το οποίο Google επανέλαβε ότι ε, θα συνεργαστεί μαζί μας και η συνεργασία αυτή είναι πραγματικά αναγκαία. Ελπίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορώ βέβαια να προκαταλάβω ε, την λύση που θα δοθεί, αλλά αναλαμβάνω τη δέσμευση και ενώπιον σας και ενώπιον των πολιτών, άλλωστε και εγώ χρησιμοποιώ το Google καθημερινά πολλές φορές, ότι θα φτάσουμε στο τέλος της έρευνας αυτής και θα δηλώσουμε εν τέλει εάν υπάρχουν προβλήματα, οπότε θα λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις. Εάν δεν υπάρχουν προβλήματα από την άποψη του ανταγωνισμού, πάλι θα το δηλώσουμε. Τώρα, πρόστιμα. Συμφωνώ μαζί σας ότι τα πρόστιμα πρέπει να είναι αρκετά υψηλά ώστε να έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα. Συμφωνώ επίσης και με το θέμα της νομικής ασφάλειας, την οποία έχουμε στο σύστημά μας. Έχουμε μια νομική βάση για την επιβολή προστήμων με τις αποφάσεις μας σε καρτέλ, σε υποθέσεις αντιτράστ. Έχουμε δημοσιεύσει και τις κατευθείαν γραμμές μας για τα πρόστιμα, τα κριτήρια δηλαδή που χρησιμοποιούμε για να αποφασίσουμε σε ποιο επίπεδο θα κινηθεί το πρόστιμο εφόσον επιβεβαιωθεί η παραβίαση. Ε, οι κατευθείαν αυτοί οι κανόνες είναι ε, δημόσιο κτήμα. Ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιούμε τους κανόνες αυτούς θα πρέπει να είναι ο αυστηρότερος δυνατός. Εν τέλει βέβαια το δικαστήριο έχει την τελευταία λέξη. Τα πρόστιμά μας λοιπόν αυτή τη στιγμή ε, το ένα μέρο ζητήσει από το δικαστήριο να εκδώσει απόφαση. Όπω είπα, την τελευταία λέξη την έχει το δικαστήριο. Το σύστημά μα λοιπόν είναι καλά προστατευμένο και στέρεο από νομική απόψεω. Είναι καλό λοιπόν το σύστημα. Ορισμένοι λένε ότι επειδή θα συμπεριλάβουμε την συνθήκη ανθρώπινων δικαιωμάτων του Στρασβούργου δηλαδή στο νομικό μας πλαίσιο αυτό ενδέχεται να προκαλέσει αλλαγές εγώ δεν συμφωνώ με τη γνώμη αυτή θα διατηρήσουμε το σύστημά μας έστω και συμπεριλαμβάνοντας την συνθήκη αυτή και το διοικητικό μας σύστημα και την πολιτική μας για τα πρόστιμα συνήθως έχουμε την ικανοποίηση να μας υποστηρίζει εν τέλει με τις αποφάσεις του το δικαστήριο και βεβαίως ε, έχουμε απόλυτο σεβασμό απέναντι στο δικαστήριο αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, συλλογικές ε, αγωγές αποζημιώσεων κλπ. Από την πρώτη μας ακρόαση εδώ, τον Ιανουάριο, ανακοινώσαμε ότι οι τρεις επίτροποι που συνδέονται περισσότερο, δηλαδή η Vivian Redding δικαιοσύνης, John Bias, προστασία καταναλωτών και εγώ προσωπικά αρμόδιος για τον ε, ανταγωνισμό, ανακοινώσαμε στο Κοινοβούλιο ότι θα θέλουμε από το Σώμα των Επιτρόπων μια συνολική προσέγγιση που δεν είναι εύκολη βέβαια, είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται και καλύτερο συντονισμός των δράσεών μας στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και πιο συνεκτική προσέγγιση, διότι οι περισσότερες διαδικασίες αναπτύσσονται ε, στα εθνικά πλαίσια, στα πλαίσια των εθνικών δικαίων δηλαδή, με διαφορετικές παραδόσεις νομικές κλπ. Κάνουμε τώρα την διαβούλευση αυτή, με τα αποτελέσματα της διαβουλεύσεως θα τοποθετηθούμε τελικά ως σώμα επιτρόπων για τις συλλογικέ αγωγές και τότε θα υποβάλω στους συναδέλφους μου και μετά στο Ευρωκοινοβούλιο την πρωτοβουλία που έχω ανακοινώσει ήδη από την ε, έναρξη της υπόθεσης αυτής των ε, συλλογικών ε, αγωγών. Δεν μπορώ ακόμα να προβλέψω ποιες θα είναι οι λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας αυτής, αλλά να είστε βέβαιοι ότι δεσμεύομαι ότι χρειάζεται να αποφύγουμε οι εσδήποτε καταχρήσεις έχουν σημειωθεί σε άλλα συστήματα και όλοι κατανοούν τι εννοώ όταν λέω άλλα συστήματα. Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα και καλώς ορίσατε. Θα ήθελα να υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις σε σχέση με την εφαρμογή της, ε, του επαναπροσδιορισμού του τραπεζικού συστήματος στην Ισπανία. Ε, ο Χωσέ Γκαρθίαντε Παλάσιος, που είναι πρόεδρος της ΚΑΧΑ, είπε ότι ορισμένες ε, τράπεζες κατέβαλαν μπόνους στους ε, εργαζόμενους. Έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα θέμα θέμη του ανταγωνισμού σε σχέση με τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και επίσης ε, μια άλλη ερώτηση. Ορισμένες τράπεζες αποτεμίευσης έλαβαν χρήματα από αυτό το σχέδιο διάσωση, ιδιαίτερα η Κάσα Καταλούνια, 1,4,8 των κονδυλίων αυτών. Άρα σε αυτή την περίπτωση τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν προσέφηγαν σε αυτόν τον μηχανισμό ε, υπόκεινται τις αρνητικές συνέπειες ενός αθέμητου ανταγωνισμού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τρεμός. Σας ήθελα να σας συγχαρώ για τα αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης Κυριακής, για το κόμμα σας. Νομίζω ότι τα ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να μπορούν να κάνουν πιστώσεις πρέπει να καταβάλουν τους μισθούς ε, στο προσωπικό. Δεν νομίζω ότι αυτό ε, αντιβαίνει, δηλαδή αντιφάσκει το ένα με το άλλο. Ως προς την αρρωγή που θα δοθεί στα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μιλάμε εδώ για δημόσιο κεφάλαιο που χορηγείται κάτω από συγκεκριμένους όρους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές. Και μέσα στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων ή ε, ε, με βάση μία ειδική διαδικασία αδειοδότησης αφορά προγράμματα που ελέγχονται από την Επιτροπή. Πρόκειται για εγγυήσεις ή υποστήριξη για αντιμετώπιση τοξικών προϊόντων ή για τη διασφάλιση ρευστότητας. Χρησιμοποιείται λοιπόν αυτή η πάγια διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, είτε στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων, δηλαδή στα μεμονωμένα προγράμματα, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλοι θα πρέπει να τηρήσουν τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που ορίστηκαν το 2008-2009. Έτσι θα συνεχίσουμε να δρούμε. Πολλές φορές ε, φαίνεται εύκολο να αποφασίζει κανείς για την ε, συμβατότητα της αρρωγής αυτής με βάση το προδιαγραμμένο πλαίσιο, άλλες φορές είναι πιο δύσκολο να οριστεί αυτό υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που συζητούνται σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δηλαδή, μια περιφερειακή τράπεζα της Γερμανίας είναι ένα ζήτημα που συζητάμε από το Μάιο του 2009 για την κατάσταση αυτής της τράπεζας, γιατί τα τοξικά προϊόντα πέρασαν σε μία άλλη τράπεζα, την επωνομαζόμενη κακή τράπεζα. Στη συνέχεια έγινε μία ε, συνάντηση με τις ομοσπονδιακές αρχές και την τράπεζα αυτή για να δούμε πώς μπορεί να γίνει μία αναδιάρθρωση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Είναι, υπάρχουν απλές περιπτώσεις και δύσκολες περιπτώσεις. Στην περίπτωση της Ισπανίας, στο ισπανικό ε, πρόγραμμα, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Τώρα, αν υπάρχουν ε, ισχυρισμοί μη συμμόρφωσης, τότε αυτό είναι διαφορετικό. Όταν αποφασιστούν αυτά τα σχέδια από τις αρμόδιες Ισπανικές αρχές. Οι Ισπανικές αρχές θα πρέπει να εγγυηθούν την τήρηση των όρων τη στιγμή που πρόκειται για μεμονωμένα σχέδια, τα οποία βεβαίως αναλύει η Κομισιόν. θα ήθελα να σας πω ότι ως προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπάρχουν δυσκολίες, αλλά οι δυσκολίες ήταν ίσονος σημασίας, συγκρίνοντας με άλλες που ισχύουν σε άλλα κράτη-μέλη. Καταφέραμε να φτάσουμε σε μία συνεννόηση με τις Ισπανικές Αρχές ως προς τα μεμονωμένα προγράμματα. Η Σόφη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ Επίτροπε για την ε, εισήγησή σας. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα δεν είχα κακή διάθεση, αλλά αφού άκουσα τα σχέδιά σας, βελτιώθηκε η κατάστασή μου και η διάθεσή μου ιδιαίτερα μετά την έρευνα ως προς το Google και υποθέσεις που σχετίζονται με το Google. Η Google μας παρέχει υπηρεσίες που δεν είχαμε ποτέ πριν, αλλά είναι γεγονός ότι το σώμα αυτό είχε εκφράσει ανησυχίες για τη δεσπόζουσα θέση της Google. Εγώ είχα οργανώσει ε, ένα σεμινάριο για τις υποθέσεις double click της Google και ζητήσαμε να ε, δούμε τι γίνεται με τη διαφήμιση στις μηχανές αναζήτησης. Η έκθεση θα ψηφιστεί αύριο το πρωί, όπως γνωρίζετε. Ε, γνωρίζω ότι δεν μπορείτε να μας πείτε τίποτα για την υπόθεση Google, γιατί δεν ξέρετε πώς θα εξελιχθεί. Θα ήθελα όμως ορισμένες διασαφήσεις από εσάς. Με εκπλήσει το ότι η διαδικασία είναι ιδιαίτερα αργή. Δηλαδή αντιδράσατε μετά από καταγγελία. Η καταγγελία υποβλήθηκε το Φεβρουάριο του 2010, δηλαδή 9-10 μήνες πριν. Και μας λέτε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας οδηγήσουν να πιστεύουμε ότι υπάρχει, γίνεται κάποιο σφάλμα. Αλλά αν σας χρειάστηκαν 9-10 μήνες να δείτε την καταγγελία, τότε θα πρέπει να έχετε σχηματίσει μία άποψη. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πόσο θέλετε να σκάψετε αυτή την υπόθεση. Στην περίπτωση της Google διπλό κλικ υπήρξε στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EFTC στη ΣΥΠΑ. Γνωρίζω ότι είναι ευρωπαϊκή υπόθεση και οι καταγγέλλοντες είναι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά είμαι σίγουρος ότι μιλήσατε με τους ομολόγους σας της ΕΠΑ. Και επαναλαμβάνω το ίδιο ερώτημα. Η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να το δει ευρύτερα το ζήτημα, δηλαδή να μην βασίζεται σε μία καταγγελία, αλλά να προβεί σε μία έρευνα του τομέα. Χρειαζόμαστε επιχειρήσεις όπως η Google, αλλά χρειαζόμαστε και ανταγωνισμό, διότι οι μηχανές αναζήτησης αποτελούν ε, βασικό αγαθό, βασική ανάγκη, είναι σαν το νερό και τον ηλεκτρισμό τις χρειαζόμαστε και δεν μπορεί να υπάρχει ένας παίκτη ο οποίος να κατέχει δεσπόζουσα θέση όπως η Google. Όσο καλή και να είναι ως μηχανή αναζήτησης, δεν μπορεί να υπάρχει αποκλειστική χρήση σε αυτές τις πρώτες ύλε όπως τις αποκαλούμε. Σας ευχαριστώ. Κατανοώ ότι θεωρήσατε ότι η αντίδρασή μας ήταν βραδύτατη στις καταγγελίες. Ίσως θα έπρεπε να είχαμε αντιδράσει, όχι επειδή ανέκυψε μία καταγγελία, αλλά επειδή ξέρουμε πώς λειτουργεί η Google ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Άρα εκ των προτέρων, μάλλον αυτεπαγγέλτος, εξοφίτιο θα έπρεπε να δράσουμε. Είναι πολύ απλό το κλικ στο Google. Δεν είναι όμως εύκολο να κατανοήσει κανείς γιατί όταν κάνει κλικ λαμβάνει ορισμένες πληροφορίες και δεν λαμβάνει άλλες. Δεν είμαι εμπειρογνώμων, δεν είμαι γνώστης, αλλά μπορώ να σας πω ότι όταν ακούω τους εμπειρογνώμονες καταλαβαίνω ότι το θέμα δεν είναι καθόλου απλό. Και δεν είναι απλό να φτάσουμε σε συμπεράσματα ότι υπάρχει παραβίαση ή παράβαση και ότι, ή ότι δεν υφίστανται προβλήματα. Γι' αυτό ανοίξαμε και την έρευνα. Έχουμε λάβει πολλές πληροφορίες, πληθώρα πληροφοριών από τους καταγγέλλοντες και από την επιχείρηση και τώρα που επίσημα έχουμε, ε, έχει ανοίξει η διαδικασία Ίσως λάβουμε περισσότερες πληροφορίες από άλλους εμπλεκόμενους φορείς που θα συνεργαστούν μαζί μας. Το ελπίζω. Τώρα, πόσο θέλουμε να σκάψουμε ε, σε αυτή την υπόθεση μέχρι τελικής πτώσεως. Αλλά πολλές φορές αυτό δεν είναι συμβατό. Δηλαδή αυτή η θέληση του να κινηθεί κανείς μέχρι τέλους και να κλείσει την υπόθεση με μία απόφαση, αυτό δηλαδή μάλλον απέχει πόρο το ένα από το άλλο. Είναι δύσκολη αυτή η διαφορά. Θα της προσδώσουμε μεγάλη σημασία και πόρους, αλλά δεν είναι η μόνη περίπτωση που μας απασχολεί. Στον κατάλογο ε, όλων των οικονομικών τομέων όπου υπάρχουν προβλήματα ανταγωνισμού. Ιδιαίτερα σε σχέση με τον καινοτόμο ψηφιακό κόσμο και δραστηριότητες. Γνωρίζουμε ότι ορισμένες εθνικές αρχές ανταγωνισμού ξεκίνησαν τις έρευνες ή βρίσκονται σε προερευνητικό στάδιο και θα συλλέξουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Ήρθαμε σε επαφή και θα συνεχίσουμε με τους ε, ε, ομόλογους των ΙΠΑ με τις αρμόδιες αρχές περί ανταγωνισμού μέσα στα πλαίσια των κανόνων απορρίτου. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τις ε, πόρτες μας και να δείξουμε όλα, όλους τους δικούς μας φακέλους ή υποθέσεις. Ελπίζω να μην χρειαστεί να φτάσουν τουλάχιστον μέχρι την δική μου γενική διεύθυνση. Και ελπίζω οι Βίκυλοι, τα Wikileaks να μην φτάσουν στη δική μου πόρτα και με καταγγείλουνε. Αλλά όταν έχετε να κάνετε με μεμονωμένες επιχειρήσεις, θα πρέπει να δούμε, να, μάλλον να τα κάνουμε όλα αυτά μέσα στα πλαίσια του σεβασμού και της στήρησης κανόνων, όταν ζητάμε συγκεκριμένες ε, πληροφορίες. Πρόκειται για νέες υπηρεσίες πολύ χρήσιμες. Ανοίγουμε νέες οδούς ευκαιριών και δυνατοντήτων, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Google κατέχει το μερίδιο του λέοντος, δηλαδή άνω του 90% στην αγορά. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης για να προωθήσουμε αυτή την έρευνα η οποία ξεκινάει από σήμερα. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριος Λάνγκεν. Ευχαριστώ. Κύριε πίτροπε. πρώτα τα συγχαρητήρια. Μετά από μια πενταετία μιας πολιτικής ανταγωνισμού που κυρίως απευθύνθηκε στον τύπο, αρχίζετε τώρα να περνάτε στην ουσία. Συγχαρητήρια. Ειλικρινά, διότι τα καλύτερα επιτεύγματα την ανταγωνιστική πολιτική θα προκύψουν εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλάβει τις ευθύνες της μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της με κάθε γαλήνη και ησυχία. Για το θέμα τώρα των οικονομικών ενισχύσεων προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα, θυμούμε ότι στις εποχές της Επιτρόπου Κρόες χρειάστηκαν 24 ώρες μέχρι να κλείσει το θέμα των ε, ενισχύσεων στις ε, τράπεζες Benelux. Τώρα εσείς έχετε κληρονομήσει μερικές παλαιές υποθέσεις όπως ορισμένων γερμανικών τραπεζών. Της Landesbank West για παράδειγμα. Εμένα με ενδιαφέρει, εδώ και χρόνια έχω τον φόβο ότι από την δική σας γενική διεύθυνση και σχετικά με αυτές τις παράπλευρες δραστηριότητες πάει να γίνει μια αναδιάρθρωση του γερμανικού τραπεζικού τομέα και κυρίως με τον στόχο να απομακρυνθούν από την αγορά οι γερμανικές Landesbank. Πώς βλέπετε λοιπόν την West LB, την ε, Landesbank West, πώς βλέπετε την υπόθεση αυτή και θα ήθελα επίσης να μου εξηγήσετε πώς κρίνεται συνολικά το θέμα των κρατικών ενισχύσεων για τον τομέα της σταθεροποίησης των τραπεζών. Ο κύριος Αλμούνια. Ευχαριστώ κύριε Ράγκεν. Πώς βλέπω και τι κάνω για τις Landesbanken. Για την ώρα έχουμε τρεις υποθέσεις, τρία σχέδια αναδιαρθρώσεως για τρεις Landesbank που τα διαπραγματευόμαστε. στην περίοδο της Νέλη Κρούς είχαμε τότε την υπόθεση της Landesbank, περιφερειακής τράπεζας δηλαδή της Βάδης Βιρτεμβέργης με ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης ακόμα διαπραγματευόμαστε τώρα της Βαβαρίας την Nord και την West του Βορρά και της Δύσης δεν μπορώ να προβλέψω πότε θα τελειώσουν οι υποθέσεις αυτό, αυτές. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι τρεις αυτές υποθέσεις είναι διαφορετικές. Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που είναι οι ίδιες, αλλά κάθε μια από τις υποθέσεις είναι διαφορετική. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα στο Αμβούργο και συναντήθηκα με τις αρχές του Ομοσπονδού Αυτοκρατηδίου και με τον Υπουργό οικονομικών του κρατηδίου Σλέσβικ Χολστάιν, που είναι και μέτοχος στην τράπεζα αυτή, για να συζητήσουμε τις υποθέσεις αυτές. Σε άλλες περιπτώσεις, συναντήθηκα με τις βαβαρικές αρχές, αλλά και με τις ομοσπονδιακές αρχές, για να συζητήσουμε την αναδιάρθρωση της βαβαρικής Landesbank. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο αναδιαρθρώσεως που θα μας ασφαλίζει τα τρία πράγματα που ζητούμε και σε όλες τις υποθέσεις αυτές. Πρώτον, ότι το σχέδιο αναδιαρθρώσεως δεν θα στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, πέραν των ορίων που είναι απολύτως βέβαια αναγκαία όταν μπαίνουν στη μέση κρατικά ε, χρήματα και ότι η τράπεζα μετά από την αναδιάρθρωση είναι βιώσιμη μέσο και μακροπρόθεσμα. Ελπίζω ότι θα ε, μπορέσουμε να ικανοποιηθούμε σε αυτές τις απαιτήσει όταν διαπραγματευόμαστε με τις περιφερειακές αυτές αρχές. Η West Bank είναι η πιο δύσκολη περίπτωση. Υπήρξε, υπήρξε μια πρώτη απόφαση τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Μετά υπήρξε μια μεταφορά τοξικών ε, στοιχείων, τοξικών δανείων 77 δισεκατομμυρίων περίπου και σύμφωνα με τους υπολογισμού μας αυτό σημαίνει ότι δόθηκαν κρατικές ενισχύσεις της τάξης των 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ίσως χρειαστεί πρόσθετη αναδιάρθρωση ή επανακαταβολή, επιστροφή δηλαδή. Μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει καμία εξασφάλιση ούτε για την ενδεχόμενη επιστροφή ούτε για την αδιάρθρωση. Τέλος, στην τελευταία μου συνάντηση με, όλες, με όλα τα ε, αναμειγνώμενα επίπεδα και τον ίδιο τον κύριο Σόιπλε και τον ε, Υπουργό της ε, Βόρειας Ινανίας της καταλήξαμε σε μια προθεσμία. Πριν από τις 15 Φεβρουαρίου θα πρέπει να υποβληθεί το σχέδιο αναδιαρθρώσεως και στείλαμε στις γερμανικές αρχές επιστολή που λέμε ποια πράγματα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο αναδιαθρώσεως. Ελπίζω μετά από αυτά τα βήματα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Πάντως, αυτές οι εξηγήσει δίνουν το μήνυμα ότι υπάρχει το πρόβλημα σε διάφορες περιφερειακές τράπεζες, Landesbank, αλλά δεν ασχολούμαστε με τον τομέα στο σύνολό του, αλλά με επιμέρους τραπεζικά ιδρύματα γιατί κάθε μία από αυτές τις τράπεζες έχουν και διαφορετικά business model. Δεν ακολουθούν όλες το ίδιο. Εγώ ορισμένα από αυτά τα business model τα θεωρώ απολύτως βιώσιμα, αλλά θεωρώ ότι θα χρειαστούν κάποιες αλλαγές για να γίνουν βιώσιμα. Φίλιπ. Είπατε και σε άλλους τομείς ότι θα μας αναφέρετε τι θα κάνετε ε, και πώς θα αντιμετωπίσετε τους ε, τομείς μελλοντικά. Ως προς το παρελθόν για τον χρηματοπιστωτικό τομέα μας είπατε ότι θα υπάρχουν ε, βασικά ενισχύσεις, βασικές ενισχύσεις για το 2011. Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα επιδοθούν το πρώτο τρίμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 2011. Και θα δούμε τις άμεσες ενισχύσεις αλλά και την επιστροφή των δανείων αυτών στον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα γίνει και η επιστροφή των ενισχύσεων, των επιδοτήσεων. Δηλαδή να αναλύσουμε ολόκληρο τον κύκλο των μετρών που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Τώρα, στρεφόμενος προς το μέλλον, Ας υποθέσουμε ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει ένα ειδικό βάρος στην πολιτική ανταγωνισμού, διότι η κρίση οδήγησε σε μία ακόμα μεγαλύτερη ε, συγκεντρωτική πορεία αυτού του τομέα, όπου λόγω μεγέθους ορισμένα ιδρύματα επιβάλλουν τους νόμους τους. Αυτή είναι η δύναμη της αγοράς και ιδιαίτερα ως προς τα στοιχεία ενεργητικού ε, γίνεται ε, στρέβλωση, δηλαδή στρέφονται από τα χρηματιστήρια στις εσωτερικές αγορές. Άρα από το ίδιο τους το βάρος ελέγχουν τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. Άρα θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα μέτρα που προτίθεστε να λάβετε γιατί ο συνάδελφός σας, ο κύριος Μπαρνιέ, και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά αυτό το τομέα. Πώς θα μπορέσετε λοιπόν να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι πολύ μεγάλες. Δεν θα πτωχέσουν αλλά και ελέγχουν την αγορά. Μία άλλη μορφή ανταγωνισμού που είναι δύσκολο να καταστήλουμε είναι η εξής. Η βιομηχανία του χρηματοπιστωτικού τομέα βρίσκεται σε ανταγωνισμό με όλες τις άλλες βιομηχανίες για να προσελκύσει κεφάλαια. Και λόγω της θέσης της προτείνει και υπόσχεται αποδόσεις που ένας ε, κατασκευαστής επίπλων, ε, ένας ε, αντιπρόσωπος αυτοκινήτων δεν μπορεί να προσδώσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις. Άρα η βιομηχανία του χρηματοπιστωτικού τομέα δεν δημιουργεί μία αξία αφεαυτής. Θεωρείτε ότι πρόκειται θέμα ανταγωνισμού και αν ναι, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ξέρω ότι το θέμα δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είσαστε και όποιος και όποιος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως προς το πρώτο ε, μέρος της ερώτησής σας για την έκθεση που σας προανακοίνωσα Ελπίζω να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία μέχρι τα τέλη Ιουνίου, αλλά δεν μπορώ να προτρέξω. Δεν ε, μπορώ να έχω έτοιμη μια τέτοια έκθεση μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, γιατί θέλουμε να συμπεριληφθούν όλες οι πτυχές. Ποιες ήταν οι επιδοτήσεις πού επιδόθηκε αυτή η βοήθεια, ποια χρήση έγινε, τι χρήση έγινε από ποιους φορείς και ιδρύματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αποτελεσματικότητα το, της χρήσης του δημόσιου χρήματος. Εδώ πολλά θα υποθούν από εκείνους που κάνουν μεταφορά χρημάτων. Εμείς θέλουμε να ελέγξουμε το πώς δαπανήθηκαν ή μεταφέρθηκαν τα χρήματα, αλλά ως προς την αποτελεσματικότητα χρήσης του δημόσιου χρήματος, δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε όλες τις πληροφορίες σε κάθε κράτος μέλος. Ή με βάση την ανάλυση που θα κάνουν τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, κατά πόσο περνάμε από τον κρατικό έλεγχο στον ευρωπαϊκό. Θα το δούμε. Ως προς συγκέντρωση δραστηριοτήτων είναι γεγονός ότι η τραπεζική δραστηριότητα υπόκειται αυστηρότερες ε, ρυθμίσεις και ελέγχους και σε ορισμένες, ως προς αποφάσεις που είχαμε λάβει πριν από την κρίση, είχαμε αποκεντρώσει ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες με το MIFID και με άλλα μέσα. Μπορούμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις να δούμε μία συγκέντρωση χρηματοοικονομικής δραστηριότητας η οποία βρίσκεται εκτός ε, ε, τράπεζας δηλαδή στον μη τραπεζικό τομέα. Ξέρουμε λοιπόν και βλέπουμε τι συμβαίνει κάθε μέρα στις οικονομικές δραστηριότητες και θα δούμε τι θα γίνει και με την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Αυτό μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι ο εξωτραπεζικός τομέας ο οποίος χρήζει περαιτέρω ανάλυσης από πλευράς ε, ρύθμισης και από πλευράς ε, της αρμόδιας για τον ανταγωνισμό αρχής. Δεν μπορώ να σας πω ότι ε, διενεργούμε μία έρευνα, όμως αυτό το τομέα θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και από πλευράς ρύθμισης και από πλευράς ανταγωνισμού. Ένα άλλο ζήτημα που θίξατε αφορά τον ανταγωνισμό για να προσελκύσουμε κεφάλαια. Ο ανταγωνισμός σε αυτή την περίπτωση είναι θετικός, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά κεφαλαίου στην αγορά. Αυτό καταρχήν δεν είναι αρνητικό. Το ζήτημα είναι ποιος θα είναι ο πλέον ανταγωνιστικός και ποιος θα ε, αποκτήσει το μεγαλύτερο μερίδιο κεφαλαίων. Όταν συγκρίναμε το ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα με το αμερικανικό, είδαμε ότι στις ΗΠΑ, στον αγγλοσαξονικό κόσμο γενικότερα και στις ΗΠΑ ειδικότερα, τα τρία, τέσσερα, τρία τέταρτα συγγνώμη, των χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων περνάνε από την κεφαλουχική αγορά ενώ στην Ευρώπη, στην υπηρετική Ευρώπη, αφορά ένα 25%. Ενώ τα τρία τέταρτα διαβιβάζονται μέσω τραπεζικού τομέα. Τώρα, ποιο θα είναι το δίκτυο διανομής στο μέλλον, θα το δούμε, γιατί θα έχουμε την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, την οδηγία κεφαλαιουχικών απαιτήσεων και ούτω καθεξής. Γι' αυτό Θεωρούμε ότι με βάση αυτή την οδηγία υπαριθμών 4 κεφαλαιοχικών απαιτήσεων θα έχουμε μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς κεφαλαίου που θα ορίζει τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Δηλαδή θα μειώσουμε την εξάρτησή μας από την τραπεζική πίστη. Αυτή θα είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Τώρα, ποιος θα μπορέσει να προσελκύσει τα κεφάλαια, αυτό είναι πολύ πρόωρο να απαντηθεί. Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στην ε, κεφαλιουχική αγορά υπό ανταγωνιστικούς όρους, τουλάχιστον επί του παρόντος. Η Βίκη. Ευχαριστώ πολύ. Μια πολύ γρήγορη ερώτηση. Θα συμφωνήσετε φαντάζομαι ότι η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. θα πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε ε, οι δικές μας οι νομοθετικές διατάξεις να ε, παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό ουσιαστικά. τους χάρη στο τομέα των αυτοκινήτων είναι πολύ δύσκολο εκεί για κάποια εταιρεία να, μετα, να μεταφερθεί από το ένα τμήμα της αγοράς σε ένα άλλο και αυτό παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό. Κάτι τέτοιο πώς μπορεί να αποφευθεί στο μέλλον και μπορούμε να βασιστούμε σε εσά κύριε Επίτροπε ο οποίο θα υποστηρίξει μέχρι τη τελευταία ρανίδο τον ανταγωνισμό. Βεβαίω, λέει ο κύριο Σαλμούνια είμαι υπεύθυνο για τον ανταγωνισμό είναι και ε, ύψιστη προτεραιότητά μου βεβαίως να πίσω τους ε, συναδέλφους επιτρόπους ότι όλες οι αποφάσεις που παίρνουμε στο σώμα των επιτρόπων πρέπει να είναι σύμμορφες με τον θεμητό ανταγωνισμό. Σε τελευταία ανάλυση όμως, όταν μιλάμε για την νομοθετική δουλειά, εσείς είστε η νομοθετική δουλειά, εσείς έχετε την εξουσία. Εάν οι προδικές σας οι προτάσεις δεν είναι 100% σύμμορφες με τον θεμητό ανταγωνισμό, ποιος φταίει. Ναι, πολλές φορές αργότερα βλέπουμε, παίρνουμε είδηση ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος, οπότε εκεί θέλουμε τη βοήθειά σας. Βεβαίως θα την έχετε, λέει ο κύριος Σαλμούνια. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα που θεωρώ άμεσου ενδιαφέροντος σε σχέση με τις κυρώσεις στον ιδιωτικό τομέα. Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία συναπόφασης και επίσης είπαμε ότι θα πρέπει αμελητοί να εφαρμοστούν. Θα θέλαμε λοιπόν να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα για αυτές. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα στο οποίο δεν αναφερθήκαμε. Ο πρώην Επίτροπος Μόντι είχε συντάξει μία έκθεση για την ε, εσωτερική αγορά και μίλησε και για, την και για τον αθέμητο φορολογικό ανταγωνισμό θα πρέπει να τηρήσουμε τις υγιείς αρχές ανταγωνισμού. Τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με μία συναγόμενη, με μία συγκαλυμμένη, ε, έναν συγκαλυμμένο προστατευτισμό μέσω επιτοκίων και μέσω άλλων μέσων. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούμε να ε, ενοποιήσουμε το φορολογικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη, διότι σε μία αγορά online πολλές οι υπηρεσίες μπορούν να συγκεντρωθούν σε μία χώρα, όπου για παράδειγμα υπάρχουν πολύ χαμηλά επιτόκια και όπου υπάρχουν ειδικέ ρυθμίσεις. Πώς ε, θα αντιμετωπίσετε ένα παρόμοιο θέμα ως προς το χρονοδιάγραμμα για τη μελλοντική πρωτοβουλία για τον ιδιωτικό τομέα και σε σχέση με τις συλλογικέ αγωγές νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μια συμφωνία στο Διευθυντήριο για τις συλλογικές αγωγές οι οποίες δεν αφορούν μόνο τον ιδιωτικό τομέα αλλά και άλλους τομείς, δηλαδή την προστασία του καταναλωτή, το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Γιατί εάν δεν υπάρχει μία συνεκτική αντιμετώπιση του θέματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και τη στιγμή που μιλάμε για συλλογικές προσφυγές ή αγωγές που δεν θα οδηγήσουν σε αυτά αποτελέσματα, τότε δεν θα φτάσουμε πουθενά. Αυτή η προγενέστερη συμφωνία είναι ύψη της σημασίας. Έχουμε ήδη προχωρήσει αρκετά. Υπάρχει δημόσιος διάλογος και θα δούμε τι θα ανακύψει έτσι ώστε το επόμενο έτος να φτάσουμε σε μία κοινή θέση, αλλά δεν μπορώ να σας πω πότε θα φτάσουμε σε αυτή την κοινή θέση, διότι δεν εξαρτάται από μένα, αλλά από το Σώμα των Επιτρόπων, από τους 26 άλλους συναδέλφους μου. Νομίζω όμως ότι δεν θα υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες για να προετοιμάσουμε το τελικό σχέδιο της πρότασης οδηγίας σε σχέση με τις συλλογικές αγωγές ή προσφυγές. Όμως δεν μπορώ να σας ε, μιλήσω για μια συγκεκριμένη ημερομηνία, διότι δεν εξαρτάται από εμένα μόνο. Εξαρτάται και από την συνεργασία με το Κοινοβούλιο εδώ και αρκετά χρόνια. Ως προς το δεύτερο θέμα που θίξατε, σε σχέση με τον αθέμητο φορολογικό ανταγωνισμό, σίγουρα είναι ε, ένα στοιχείο που διέπει τις αγορές και επηρεάζει τις οικονομικές αποφάσεις ως προς μια επένδυση σε ένα σημείο της Υπήρου ή την μετεγκατάσταση μιας επιχείρησης στην εσωτερική αγορά. Υπάρχουν όμως δύο στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ούτε η Επιτροπή ούτε το Κοινοβούλιο. Καταρχήν, σύμφωνα με την ε, πάγια νομολογία μας, ο φορολογικός ανταγωνισμός θα πρέπει να τύχει έρευνας, δηλαδή να δούμε ποιες είναι οι παραβάσεις ε, μέσα σε κάθε κράτος μέλος. Δεν μπορούμε να είμαστε επιλεκτικοί. Γιατί θα πρέπει να δούμε πώς δρούν οι οικονομικοί φορείς κάτω από ίσες και δίκαιες συνθήκες, γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να την χάνουν ίσες μεταχείρισης ως προς την φορολόγηση στα κράτη-μέλη. Και πέρα από τις εθνικές ε, φορολογικές νομοθεσίες θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχουν ε, ειδικά, ειδικοί φόροι, έμεση φόροι, ή επαναπροσδιορισμός ή μεταφορά κεφαλαίων. Μπορεί λοιπόν κανείς να προβάλλει ε, βέτο, διότι πρέπει να υπάρχει ομοφωνία σε φορολογικά ζητήματα ως προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Αυτό ισχύει. Ε, νομίζω ότι οι θέσεις μας συμπίπτουν για το τι θα κάναμε με αυτή την ομοφωνία ως προς το θέμα αυτής της ομοφωνίας που έχει εγγραφεί στη συνθήκη βεβαίως. Ο, ο Βολφ Κλίντς, κύριε Επίτροπε, με ενδιαφέρει μετά από μια συγχώνευση πώς εξετάζεται εάν οι αρχικές σας υποθέσεις ότι η συγχώνευση δεν οδηγεί σε μονοπωλιακές δομές, τουλάχιστον σε επιμέρους τομείς. Τι είδους συστημική ανάλυση κάνετε για να μπορείτε να αντιδράσετε. Συγκεκριμένο παράδειγμα. Στις, ε, έρχομαι συνήθως από τη Φραγκφούρτη με το αεροπλάνο. Μέχρι πριν από 2-3 χρόνια ήταν δύο γραμμές, η Φραγκφούρτη και η Essen Brussels η Brussels Airways, συγγνώμη. Από τότε όμω που αγοράστηκε η Brussels Airways από τη Lufthansa, οι τιμές ανέβηκαν κατά 50%, οι ε, υπηρεσίες είναι λιγότερο καλές, λιγότερες οι συνδέσει, οι πτήσει δηλαδή, κατά τη γνώμη μου πρόκειται για σαφέστατη de facto μονοπωλιακή θέση στη γραμμή Βρυξέλλες-Φραγκφούρτη. Δεν νομίζω να το έχει ε, αντιληφθεί αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ισχύ σας να εγγύψετε στο θέμα αυτό, σας προσκαλώ. Τώρα για το δεύτερο, η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν έγινε αυτό όλοι υποθέσαμε ότι θα προκύψουν μειώσει των τιμών όπως είδαμε και στις τηλεπικοινωνίες. Χρόνο με το χρόνο διαπιστώνουμε ακριβώς το αντίθετο. Τώρα περί τα τέλη του έτους λαμβάνουμε τουλάχιστον στη δική μου χώρα λαμβάνουν όλοι επιστολές για το ρεύμα, για το φυσικό αέριο κλπ. που μας λένε λίγο πολύ το ίδιο. Από 1η Ιανουαρίου δυστυχώς θα αυξήσουμε τις τιμές μας και τα ποσοστά είναι διψήφια. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι πάλι εκεί de facto υπάρχει ένα ολιγοπόλιο το οποίο χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που του προσφέρει η θέση αυτή συστηματικά για να αυξάνει τις τιμές ο Επίτροπος. Σας ευχαριστώ κύριε Κλίντς. Σε αυτό το δρομολόγιο, Φραγκφούρτης Βρυξέλλες, με επιστροφή, όταν ήμουν ε, Επίτροπος Οικονομικών, πήγαινα συχνά. Και μάλιστα και πριν από λίγες μέρες, μετά από δική σας πρόσκληση, πήρα το αεροπλάνο στο δρομολόγιο αυτό. Θα το εξετάσω. Θα το εξετάσω αυτό που μου είπατε. Μου δώσατε μια καλή ιδέα. Δεν ξέρω αν θέλετε να υποβάλλετε επίσημη καταγγελία. Οπότε θα την εξετάσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, όπως είπα στην αρχική μου ομιλία, στην εισαγωγική μου ομιλία, ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο του 2007 μια έρευνα κατά τομέα που μας απέδωσε πολλές ιδέες και υπό την ρυθμιστική μας ιδιότητα ορισμένες ρυθμίσεις που έχουν υποβάλει οι συνάδελφοί μου που είναι αρμόδιοι για την ενέργεια βασίστηκαν σε αυτή την έρευνα του τομέα που έγινε τότε. Άνοιξε και ένας κατάλογος, μια λίστα υποθέσεων από μας ως αρμοδίων ε, επί της ε, ε, επί της πολιτικής ανταγωνισμού. Εξακολουθούμε και έχουμε ανοιχτές πολλές υποθέσεις. Αναλύουμε, για παράδειγμα, τα ε, τιμολόγια των εταιριών ηλεκτρικού, επίσης φυσικού αερίου. Είμαστε πολύ απασχολημένοι και σε ορισμένα μάλιστα, σε ορισμένες μάλιστα ε, περιπτώσεις έχουμε λάβει και αποφάσεις σχετικά με ε, την ε, κατάργηση εμποδίων στην πρόσβαση, για την κατάργηση δεσπόζητας θέσης κλπ. Κατάχρηση μάλλον θέσης κλπ. Δυστυχώς οι τιμές της ενέργειας δεν εξαρτώνται μοναχά από τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση των τιμών. Στο, όταν μίλησα για antitrust είπα τέσσερις τομείς. ICT, μίλησα για το Google, πληρωμές με τις ε, πιστοτικές και χρεωστικές κάρτες μεταξύ άλλων, τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, θα μπορούσα να πω και άλλους τομείς. Και μίλησα και για την ενέργεια που είναι τομέα κλειδί και εργαζόμαστε πραγματικά πολύ σκληρά και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά στον τομέα αυτό. Και αν ε, χρειαστεί θα ζητήσω την υποστήριξη της Επιτροπής Οικονομικών της Ευρωβουλής γιατί όπως γνωρίζετε σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και κάποια διάδραση μεταξύ δημόσιας πίεσης και ιδιωτικών συμφερόντων στον τομέα αυτό και από την άποψη τη πολιτική αντιτράστη δεν είναι και εύκολο ο τομέας αυτό. Πάντως εμεί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Έχω βάλει και το όνομά μου στη λίστα των ερωτώντων και άλλωστε ο κύριο Λάγκεν θέλει να επανέλθει Μου έκανε εντύπωση που αναφερθήκατε στη σωστή διαδικασία κατά την αρχική σας ομιλία. Χαίρομαι που είπατε ότι θα υποστηρίξετε τα δικαιώματα των επιχειρήσεων, θα καταβάλλετε πάσα προσπάθεια για να μπορέσετε να γίνουν σεβαστά κάποια δικαιώματα και ότι θα φροντίστε να μην ε, επαναληφθούν κάποια πράγματα που έγιναν στο παρελθόν όπου φαινόταν ότι κάποιοι δυσαρεστούνταν αν ας πούμε μια επιχείρηση ε, το δικαίωμά της για έφεση κτλ. Τέλος πάντων και μιλάτε για, είπατε, μιλήσατε και για ένα κώδικα δεοντολογίας που θα πρέπει να τηρείτε, ε, σωστές διαδικασίες κτλ. Εγώ θέλω να καταλάβω όμως θα φροντίστε να γίνει διάκριση μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών και αρμοδιοτήτων γιατί πολλές φορές η Κομισιόν είναι τελικά και ο ανακριτής και ο δικαστής ξέρετε σε κάποιες ιστορίες Επίτροπος είπα ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες κάθε φορά που θα, υπάρχει, α, θα υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι επιδάχεται βελτίωση η συγκεκριμένη διαδικασία. Το 2011 θα είπα ότι θα προτείνουμε κατά πάσα πιθανότητα μετά τις διαβουλεύσεις και μετά τις συζητήσεις που θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα θα υποβάλουμε λοιπόν προτάσεις για τις βέλτιστες πρακτικές για να βελτιώσουμε τη διαφάνεια, για να βελτιώσουμε την τήρηση των δικαιωμάτων των διαδίκων, για να ήδη ε, προσλάβαμε ένα καινούριο άτομο πολύ ικανό για να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά είμαστε ανοιχτοί και νομίζω ότι δείχνουμε ότι είμαστε και ανοιχτοί για να βελτιώσουμε τις διαδικασίες Ωστόσο, τους τελευταίους δέκα μήνες έχω πει επανειλημμένα και το επαναλαμβώ, δεν πρόκειται να αλλάξω το σύστημα. Γιατί το διοικητικό σύστημα που έχουμε είναι το, το ίδιο καλό όπως και άλλα συστήματα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι το καλύτερο σύστημα, αλλά τέλος πάντων αυτό μπορεί να το πιστεύουν όλοι. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Ειλικρινά πιστεύω ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημά μας, τους πυλώνες του σύστηματός μας. Το θέμα αυτό τώρα της διάκρισης και του διαχωρισμού. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι στο παρελθόν, πολύ παλιά, υπήρχε ο διαχωρισμός αυτός μέσα στην Κομισιόν. Δεν ήταν πιο αποτελεσματικό ή πιο καλό το τωρινό σύστημα. Απλώ ήταν διαφορετικό. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, είμαστε διαφανείς, έχουμε καλές σχέσεις με τους, με τους διαδίκους, ε, θέλουμε να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα αυτά τα κάνουμε πάρα πολύ καλά και το δικαστήριο επανειλημμένα έχει επιβεβαιώσει ότι το σύστημά μας συμμορφούνται με όλους εκείνους τους κανόνες με τους οποίους θα έπρεπε να συμμορφώνεται. Τώρα από εκεί και πέρα ζητώ συγγνώμη δεν είμαι 100% Αγγλοσάξον για, για το συγκεκριμένο θέμα. Έχω μια νοοτροπία έτσι εν μέρει Αγγλοσαξονική όχι πλήρως. Βέρνερ, επί, κύριε Επίτροπε, άκουσα αυτά που είπατε στον κύριο Κλίντς. Θα ήθελα κι εγώ λοιπόν να επανέλθω στο ερώτημα που ετέθη από τη συνάδελφο των πρασίνων. Ε, είναι το θέμα. Θα ήθελα να επανέλθετε σε αυτό και να μας δώσετε μερικές παραπάνω λεπτομέρειες. Excuse me, Mr. Langen, I, didn't got your... Συγγνώμη κύριε Λάγκεν, δεν κατάλαβα την ερώτησή σας. Υπάρχει μια υπόθεση στη Γερμανία που είναι το Νιονμπογκ Ρινγκ είναι ένας τόπος όπου υπάρχουν πολλές βιομηχανίες και στις οποίες δόθηκαν ειδικέ επιδοτήσεις ένα είδος κρατικής ενίσχυσης τι έχετε να πείτε γι' αυτό ε, συγγνώμη λέει ο κύριος Αλμούνια θα σας στείλω γραπτά την απάντησή μου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 Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο που ήταν εδώ. Θα σε ξαναδούμε βεβαίως το 2011 ξανά. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για το έγγραφό σας, το οποίο είναι μια σύνοψη ουσιαστικά της ομιλίας που κάνατε στην αρχή της συνάντησής μας. Μπορείτε να χειροκροτήσετε αν θέλετε, δεν απαγορεύετε. We just got a couple of minutes uh, whilst we change over and uh,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 Καθίστε πάλι παρακαλώ όλες και όλοι για να έχουμε στη διάστησή μας ε, το μέγιστο δυνατό χρονικό περιθώριο για τον ε, νομισματικό διάλογο. Καλωσορίζω και πάλι τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κύριο Ζαν claude στον τακτικό ε, νομισματικό διάλογο. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τις 27 Σεπτεμβρίου που ήταν η τελευταία φορά που τον είδαμε. Θα έχουμε ωστόσο μακρότερη περίοδο μέχρι την επόμενη φορά που θα τον δούμε στις 21 Μαρτίου. Θα ακολουθήσουμε τη συνηθισμένη διαδικασία. Θα κάνει ο πρόεδρος Τρισέ μια πρώτη τοποθέτηση και μετά θα προχωρήσουμε σε σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων. Και αν είστε όλες και όλοι φρόνιμοι, θα ακούσουμε μία ερώτηση, μία απάντηση. Thank uh, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, από την τελευταία μας συνάντηση τον Σεπτέμβριο, οι κυβερνήσεις, ζητήθηκε από τις κυβερνήσεις να δείξουν την διάθεση να σταθεροποιήσουν το ευρώ στην ζώνη ευρώ. Με το πρόγραμμα σταθεροποίησης που εγκρίθηκε από την Ιρλανδική κυβέρνηση μετά από τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διασύνδεση και με το Νομισματικό Ταμείο και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με την οπτική αυτών των εξελίξεων θα ήθελα στην εισαγωγή μου να περιοριστώ σε δύο βασικά θέματα. Την γενική οικονομική κατάσταση στην ζώνη ευρώ, καθώς και στο σχεδιαζόμενο νέο οικονομικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερος για την ζώνη ευρώ. Το σημαντικό θέμα της μεταρρύθμισης της οικονομικής διαχείρισης που γνωρίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την, για την Επιτροπή σας και θα έρθω εν τέλει και στην ε, μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού. Σε ό,τι αφορά τις μακροοικονομικές οπτικές, επιβεβαιώνεται η πεποίθησή μας ότι ανακάμπτει η ευρωπαϊκή οικονομία. Οι ρυθμοί πληθωρισμού στην ζώνη ευρώ είναι 1,9% περίπου και εκεί περίπου θα κινηθεί ο πληθωρισμός τους επόμενους μήνες πριν να μετριαστεί η πορεία του τον επόμενο χρόνο. Η, η απουσία πληθωριστικών και αντιπληθωριστικών τάσεων συνεχίζει και η προσπάθεια, σήμα, η προσπάθεια μας είναι να παραμείνει ο πληθωρισμός λίγο κάτω από το 2%. Η νομισματική μας ανάλυση επιβεβαιώνει ότι θα συνεχίσουν οι τάσεις αυτές. Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών δείχνουν ότι τα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αρχίζουν να δείχνουν πάλι αυξητικές τάσεις, ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά παραμένουν σε θετικά επίπεδα. Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση Δυστυχώς βρισκόμαστε μόλις δύο ημέρες πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την επόμενη Πέμπτη. Λοιπόν, πρέπει να σας μιλήσω για αυτή την περίοδο. Δεν μπορώ να προκαταλάβω σύμφωνα με τους κανονισμούς μας ποιε αποφάσεις θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά όπως γνωρίζετε, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ε, λαμβάνονται με στόχο να εκπληρώσουμε την εντολή μας, δηλαδή της ε, διατήρησης σταθερότητας του ευρώ. Στρεφόμενος τώρα στα θέματα που έχετε θέσει, θα πω λίγα λόγια για τις εξελίξεις των ε, συναγματικών ισοτιμιών. Η έννοια του νομισματικού πολέμου νομίζω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Δεν χρειαζόμαστε πολέμους ουδενός είδους. Χρειαζόμαστε συνεργασία μέσα σε πεποίθηση. Χρειάζεται, υπάρχουν δύο θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη σοβαρά. Πρώτον, η σχέση μεταξύ των μιζώνων ε, νομισμάτων όπως την λίρα στερλίνα, το δολάριο, το ευρώ, το γεν, το καναδικό δολάριο κλπ. Αυτά τα νομίσματα και στην περίπτωση του ευρώ και τα νομίσματα που προηγήθηκαν του ευρώ κυμαίνονται από τότε που ε, κατέρευσε στις αρχές του 70 το σύστημα Bretton Woods. Όλοι θεωρούμε ότι η υπερβολική πτυτικότητα και οι εξελίξεις των ε, συναγματικών ισοτιμιών έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομική σταθερότητα. Το δεύτερο θέμα είναι των αναπτυσσομένων οικονομιών της αγοράς με πλεονάσματα και με συναλλαγματικές ισοτιμίες που δεν είναι αρκετά εύκαμπτες έχουν αναλυφθεί τώρα δεσμεύσεις από το G20 για να προχωρήσουν σε πιο εύκαμπτες συναλλαγματικές ισοτιμίες που να επιτρέπουν και την ανατίμηση των νομισμάτων ε, των αναπτυσσομένων αυτών οικονομιών, κάτι το οποίο θα είναι προς το συμφέρον και των αναπτυσσομένων οικονομιών και της διεθνούς κοινότητας επίσης. Για την μεταρρύθμιση της οικονομικής διαχείρισης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για το M, δηλαδή για το νομισματικό, αλλά βέβαια έχουμε απόψεις και για το E, το ε δηλαδή, την οικονομική δηλαδή διαχείριση, αφού επ' αυτής εσείς εργάζεστε και αυτό με ρωτήσατε. Είχα την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα να απευθύνω το λόγο στην ε, Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και να πω ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν βελτίωση του, του πλαισίου εποπτείας για τα μέλη και εκτός, για τις χώρες μέλη και εκτός της ζώνης ευρώ. Το Συμβούλιο μας θεωρεί πάντως ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι αρκετά τολμηρά για να οδηγήσουν σε απόλυτη ε, σταθερότητα και στη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Καλύτερη λειτουργία της Οικονομικής Ένωσης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ε, σταθερότητα της ζώνης ευρώ. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν αρχίσει τώρα το νομοθετικό του έργο και αφήσει έχει γίνει αυτό, επιτρέψτε μου να έρθω στις προτινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις. Ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το προληπτικό του μέρος, οι προτάσεις της Κομισιόν κινούνται προς σωστή κατεύθυνση για ένα αριθμό θεμάτων. Συμφωνούμε καταρχήν με την προσέγγιση για σόφρονες ε, δημοσιονομικές πολιτικές, ωστόσο για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης χρειάζεται να προσθεθούν ορισμένες λεπτομέρειες και νομίζουμε επίσης ότι τα περιθώρια αποκλήσεων από σόφρονες πολιτικές δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη σημαντική ανανέωση, η αύξηση των κριτηρίων του χρέους στη βάση ε, ενός αριθμητικού benchmark είναι καταρχήν καλοδεχόμενη, αλλά μας απασχολεί το γενικώ ότι ίσως να μην είναι επαρκώς φιλόδοξο το μέτρο. Επίσης, για να εξασφαλιστεί πλήρης εφαρμογή του μέτρου, πρέπει ο χώρος ε, παρεμβάσεων να είναι πολύ περιορισμένος. Δεύτερο, για τα μέτρα επιβολής και κυρώσεων, μαζί και με ενίσχυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, το δικαίωμα υποβολή προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Αυτά πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση για ένα σχεδόν αυτόματο σύστημα. Όμως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει σημαντικέ επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά το σύστημα που ζητεί η ίδια η χώρα μέλο ή ε, σε βάση εξαιρετικών συνθήκων. Οπότε τότε μπορεί ε, οι κυρώσει αυτέ να έρονται και τότε αυτό ανοίγει σημαντικό περιθώριο ελιγμών. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει σημαντικές αμφιβολίες για τις, ε, σε περίπτωση δηλαδή οικονομικής μείωσης. Ε, είναι σημαντικό να ενισχυθούν περαιτέρω οι εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο σοφών στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να κάνει ε, εξωτερικές αξιολογήσεις των δημοσιονομικών πολιτικών και της εφαρμογής των πλαισίων. Αυτά τα μέτρα λοιπόν δεν έχουν επαρκώς αντιμετωπιστεί στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη γνώμη μας. Τέλος, οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις είναι και εθνικές δεσμεύσεις και βεβαίως εξακολουθούμε να τις ε, εξετάζουμε και μέσα στα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια με ελάχιστες προϋποθέσεις και ως ελάχιστες, και ελάχιστες προϋποθέσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι ως προς τις προβλέψεις για την φορολογική πολιτική και την ε, μεταφορά ε, αυτών των διατάξεων στο εθνικό δίκαιο. Τώρα, ως προς τις ε, μακροοικονομικές ανισορροπίες, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλήρες ε, εποπτικό πλαίσιο, ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Ζώνη που κλείνει ένα μεγάλο κοινό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την μακροοικονομική σταθερότητα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ορίσουμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες για να δούμε ποιες χώρες έχουν χάσει ε, λόγω αθέμητου ανταγωνισμού ή μη ύπαρξης ανταγωνισμού ε, λόγω και ελλημάτων. Επίσης θα πρέπει να βρούμε τους κατάλληλους δίκτες και τα κατόφλια, διαφορετικά η οποιαδήποτε συζήτηση θα, ε, δεν θα είχε κανένα νόημα. Επίσης θα πρέπει να συνδέσουμε με το βαθμολόγιο με την διαδικασία εποπτείας και μελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το ΕΚΤ για τις χώρες της Ευρωζώνης και μη. Οι κυρώσεις και άλλα μακροοικονομικά μέτρα δεν θα πρέπει να μπαίνουν αργά στη διαδικασία μετά από τη μη συμμόρφωση κρατών μελών. Θα πρέπει να ισχύουν βαθμιαία και αρκετά νωρίς για να δημιουργούν τα κατάλληλα κίνητρα. Υπάρχουν ε, κίνδυνοι οι οποίοι θα πρέπει να αρθούν. Ιδιαίτερα κάτω από έκτακτες οικονομικές συνθήκες που μπορεί να τύχουν διαφορετικής ερμηνείας. Ε, γι' αυτό θα ήθελα να είμαστε φιλόδοξοι και, έγκαιρα, και να δράσουμε έγκαιρα με αυτό το νομοθετικό πακέτο μέσα στα πλαίσια της εποπτείας για την φορολογική ενοποίηση και την εποπτεία των μακροοικονομικών ανισοτήτων. Ιδιαίτερα ως προς τα μέλη της Ευρωζώνης ως προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, Σταθερότητας, στον οποίο αναφέρθηκε την Κυριακή το Eurogroup, μετά τις 28 Οκτωβρίου ζήτησα από τις κυβερνήσεις να αποφύγουν αμφισημίες σε σχέση με επενδυτές και κατάσταση της αγοράς και τόνισα ότι η Ευρωζώνη θα πρέπει να συμβαδίζει με τις πρακτικές του Δουνουτού και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Αυτό ε, επικυρώθηκε από τις κυβερνήσεις την προηγούμενη Κυριακή. Θα ήθελα να κάνω και ορισμένα σχόλια σε θέματα του χρηματοοικονομικού τομέα. Έχετε επιτελεσθεί μεγάλη πρόοδος μετά από την αναθεώρηση της ατζέντα και τα δεδομένα των G20 και των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων νωρίτερα αυτό το μήνα. Έτσι συμμετέχουν παγκοσμίως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για να είναι πιο ανθεκτικό το χρηματοοικονομικό σύστημα. Θα ήθελα να τονίσω τρία ζητήματα. Τα πλαίσια της Βασιλείας 3, όπως εγκρίθηκαν από τους εθνικούς ρυθμιστές που αποτελεί τον ακρογωνιαίο ε, λίθο της αναθεώρησης αυτής και γι' αυτό χρειάζεται εφαρμογή και μεταφορά σε εθνικό επίπεδο. Ενώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες που θα πρέπει να συμβαδίζουν με το πλαίσιο της Βασιλείας 3 θα ήθελα να ε, τονίσω τη σημασία της μεταβατικής περίοδου ως προς την οδεία σε σχέση με την εναλλακτική επενδυτική διαχείριση θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συγκλίνουσα εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να υπάρχει δίκαιη πρόσβαση όλων των εμπλεκομένων φορέων διεθνώς. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε πρωτοβουλίες ρύθμισης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να φτάσουμε στα ευκταία αποτελέσματα χωρίς να αποτελέσουμε τροχοπέδι στην οικονομική ανάκαμψη. Σε σχέση με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, θα αρχίσουμε τον Ιανουάριο του 2011 αυτό τον συντονισμό έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτή την εποπτεία αναλύοντας τους συστημικούς κινδύνους και τις ανησυχίες όλων των εμπλεκομένων φορέων. Πιστεύω ότι αυτός ο μηχανισμός θα τεθεί σε εφαρμογή πώς προτάθηκε από το Κοινοβούλιο για να προωθήσουμε τη δυνατότητα των εθνικών και ευρωπαϊκής αρχών να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες προκλήσεις. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στα μέλη ότι έχουμε ήδη προετοιμάσει ένα κατάλογο ομιλητών. Αρχούμε, αρχίζουμε με το ΕΛΚ. Ο Ζαν Πολ Γκοζές. Γνωρίζω ότι ότι αυτές τις αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή και από τη θέση σας δεν μπορείτε να απαντήσετε εύκολα σε ορισμένες ερωτήσεις που έχουν επιπτώσει στη χρηματοπιστωτική αγορά. Θα σας υποβάλω λοιπόν τρεις ερωτήσεις που απασχολούν τους πολίτες. Έχετε μία ε, απάντηση στις επιπτώσεις ντόμινο στις αγορές. Επίσης, ως προς την αναδιάρθρωση του χρέους για μία χώρα της Ευρωζώνης, αυτό είναι ένα ερώτημα ταμπού και τι πιστεύει η ΕΚΤ ως προς τις συζητήσεις στο, στην Ευρωζώνη, ως προς την ανταγωνιστικότητα στα κράτη-μέλη. Και εδώ τελειώνει και το όνειρό μου, μαζί με την ερώτησή μου. Έχετε το δικαίωμα, το δικαίωμα να ονειρεύεστε εσεί, αλλά εγώ δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Θα ήθελα να πω το εξή. Γνωρίζετε και είσαστε μάρτυρες ε, μιας κατάστασης, γιατί εμείς βρισκόμαστε έξι φορές το χρόνο, κατά μέσο όρο αναφέρουμε ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η εποπτική αρχή, σχετική εποπτεία, είναι ύψης της ε, σημασίας για την ΟΝΕ. Υπάρχουν ευθύνες μέσα στα πλαίσια της ΟΝΕ. Η υπεύθυνοι είναι οι κυβερνήσεις και το Eurogroup είναι η ένωση των χωρών της Ευρωζώνης. Αυτό το λέγαμε από την απαρχή του ευρώ. Μετά το 2004, μάλλον το 2004, πολλές χώρες θέλαν να αποδυναμώσουν το σύμφωνο σταθερότητας και η δική σας χώρα το έκανε αυτό κύριε Γκοζές, μην το ξεχνάμε αυτό, μεταξύ των οποίων ήταν όλες οι μεγάλες χώρες που ζήτησαν την αποδυνάμωση. Εμείς είπαμε ότι ήταν ένα πολύ σοβαρό λάθος. Η ΟΝΕ χρειάζεται και τις, τους δύο πυλώνες, τον οικονομικό και τον νομισματικό. Δώσαμε μεγάλη μάχη, η Επιτροπή έδωσε μεγάλη μάχη και φτάσαμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και το δικαστήριο έδωσε μία σολομόντια λύση. Εμείς όμως γνωρίζαμε ότι βρισκόμαστε σε μία κατάσταση ρήξης. Εγώ εξ των διοικητών των τραπεζών είπα ότι είχαμε σοβαρές ανησυχίες, grave concerns είχα αναφέρει το 2005 όταν ε, φτάσαμε στο νέο σύμφωνο σταθερότητας και έκτοτε λέγαμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε την εποπτεία των δημοσιονομικών πολιτικών. Και αυτό που βλέπουμε τώρα με το ευεργέτημα του χρόνου ε, οδηγεί σε μη κατανόηση τις τάσεις του Eurogroup εκείνη την εποχή το 2004-2005. Είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να εποπτεύσουμε τους δείκτες ανταγωνιστικότητας, το ενιαίο κόστος παραγωγής και τις εθνικές ανισότητες στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Αυτό καθίστε τα απόλυτα σαφές. Οι κυβερνήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τι συνέβη και ενώπιον μιας δύσκολης κατάστασης αυτή τη στιγμή λαμβάνουν τις ευθύνες που κρίνουν σκόπιμες, οι οποίες έχουν υποτιμηθεί εν μέρη από τους παρατηρητές. Αυτό το λέω εν παρόδο. Νομίζω ότι υπάρχει η υποτίμηση των αντιδράσεων. Δηλαδή η εκτελεστική εξουσία είναι αποφασισμένη Και αυτό το βλέπουμε και από το Συμβούλιο των 27 και από το Σώμα των Επιτρόπων. Και βλέπουμε ότι δεν πρόκειται για μια νέα κατάσταση. Οι παρατηρητές δύσκολα κατανοούν τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα μπορώ να σας πω, όχι σε κατάσταση ενυπνίου, αλλά μέσα στα πλαίσια της πραγματικής κατάστασης ότι έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση διαρκούς αμφισβήτησης. Και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό θέμα. Και ως προς την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα είχα πει ότι πρέπει να οριστικοποιήσουμε, να διασαφηνίσουμε την κατάσταση, κάτι το οποίο έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οι Ευρωπαίοι διαθέτουν τους κανόνες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και κανένας Ευρωπαίος αυτή τη στιγμή δεν λέει κάτι το διαφορετικό. Διότι οι δύο χώρες που βοηθούμε έχουν, βρίσκονται σε κατάσταση φερεγγιότητας, αλλά θα πρέπει να προβούν σε προσαρμογές. Και δεν πρέπει να αμελήσουμε την σοβαρότητα αυτών των αναγκαίων προσαρμογών παντού στην Ευρώπη. Νομίζω ότι απάντησα στις δύο πρώτες ερωτήσεις σας, αλλά θα ήθελα να τις σχολιάσω περαιτέρω. Οι παρατηρητές, όπως είπα, δεν μπορούν να αποτιμήσουν αυτή την κατάσταση νέας οικοδόμησης της Ευρώπης. Υπάρχουν τέσσερα σημεία υποτίμησης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες προβαίνουν σε σταθεροποίηση και δημοσιονομική ανάκαμψη. Άλλοι βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση ως προς το σημείο εκκίνησης σε σχέση με αναπτυγμένες, άλλες αναπτυγμένες χώρες σε σχέση με τον ενοποιημένο ευρωπαϊκό χώρο. Το 2010 το, το έλλειμμα είναι 6,7% του ΑΕΠ, ενώ τον ΙΠΑ είναι 11% του ΑΕΠ. Της Ιαπωνίας 9,6% του ΑΕΠ. Αυτό για να σας δώσω ορισμένες τάξεις μεγέθους. Στην Ευρωζώνη το 2011 θα είμαστε στο 4,6% του ΑΕΠ, στις 8,9% και στην Ιαπωνία επίσης 8,9% του ΑΕΠ. Αυτό θα είναι το έλλειμμα. Αυτό δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητό. Επίσης, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει εκπλήξει και εκπλήσει διαρκώς, διότι είναι πιο δυναμική από ό,τι αρχικά προβλεπόταν μετά την ε, επαναφορά της διαδικασίας ανάπτυξης και ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης έχουν το επίπεδο Info Institute. Και αυτό το βλέπουμε το είχαμε δει και με την επανένωση της Γερμανίας που αποτελεί το 30% της Ευρωζώνης. Άρα η πραγματική οικονομία λειτουργεί στην Ευρωζώνη και εξέπληξε θετικά. Ένα τρίτο σημείο το οποίο είναι σημαντικό είναι το εξής. Το γεγονός ότι υπάρχουν μέσα και μηχανισμοί που λειτουργούν. Και αυτό το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο και το είδαμε και το προηγούμενο Κυριακό. Θα σταθώ εδώ, δεν θέλω να σας κουράσω, θα ήθελα απλώς να πω ότι και εμείς εκδίδουμε ένα νόμισμα που φέρει το όνομα ευρώ και το οποίο κράτησε την αξία του πολύ καλύτερα από τα άλλα νομίσματα την τελευταία πενταετία. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν πρέπει να υποτιμήσουμε και εμείς εκδίδουμε αυτό το νόμισμα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτά ήθελα να σας απαντήσω, κύριε Γκοζές. Ναι, ήταν ουσιώδη τα ερωτήματα και ουσιώδης και η απάντηση. Θα πρέπει να είμαστε ε, ε, λίγο πιο σύντομοι και με τις ερωτήσεις και με την απάντηση. Είμαι βεβαία ότι ε, αυτό το σεβαστείτε όλοι. Χωσέ Γκαρσία Μαργάγιο, παρακαλώ, η επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχω την υποχρέωση να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να μην μου απαντήσετε. Θα συνεχίσετε με τα έκτακτα μέτρα περί ρευστότητας το 2012. Θα συνεχίσετε να, αγορα... να αγοράζετε ε, δημόσιο χρέος το δημόσιο χρέος των κρατών. Γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφανθεί και να μας πείτε πώς θα συμμετάσχουν και οι ιδιώτες επενδυτές, ιδιωτικοί επενδυτές, μέσα στα πλαίσια της, ε, των σχεδίων διάσωσης των μελλοντικών. Το Συμβούλιο αποφάνθηκε ότι θα βλέπουμε την κατάσταση αναπερίπτωση, το οποίο σημαίνει ότι προσθέτεται στην κατάσταση αμφισημίας και αμφιβολιών που υπάρχουν και βεβαίως οι κλειδονισμοί της αγοράς συνεχίζονται κατά αυτόν τον τρόπο. Thank you very much Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όπως είπα ήδη προηγουμένως, θα εξετάσουμε την νομισματική μας πολιτική σε δύο ημέρες. Δεν μπορώ ακόμα να προκαταλάβω, όπως είναι ευνόητο, τις αποφάσεις του Συμβουλίου των Διοικητών. Και αυτό ισχύει και για την νομισματική πολιτική, αλλά και για τα άλλα στοιχεία νομισματικής πολιτικής, τα μη στάνταρτ μέτρα δηλαδή. Διευκρινίζω μόνο ότι εμείς έχουμε τα μέτρα νομισματικής πολιτικής για την εξασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και τα μη στάνταρτ μέτρα τα οποία έχουν ως σκοπό όταν χρειάζεται να βελτιώσουν τη λειτουργία των μηχανισμών μεταφοράς της νομισματικής πολιτικής όταν υπάρχουν αγορές δηλαδή οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα για το δεύτερο ερώτημα. Είπα πριν από λίγο ότι η δήλωση ήταν μια χρήσιμη διευκρίνηση διότι αναφέρεται και, στους, και στον μελλοντικό διαρκή μηχανισμό, μόνιμο μηχανισμό που θα είναι πλήρως συμμορφούμενος με τις πολιτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με τις πρακτικές του, και το λέω εδώ, το γράφω, το έχω ξαναπεί ξανά και ξανά, γιατί ένα από τα αμφίσιμα σημεία ήταν εάν θα υπάρξει νέο κόνσεπτ που δεν είναι αυτό που χρησιμοποιείται στον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό, αυτή η διαφορετική έννοια, αυτό το διαφορετικό κόνσεπτ, κάπως, για να πω ε, διπλωματικά, εκφόβησε τους επενδυτές που ανησυχούσαν για τις επενδύσεις τους στην Ευρώπη. Ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό αυτή η αμφιβολία, η αμφισημία που κράτησε περίπου ένα μήνα να διευκρινιστεί απολύτως. Νομίζω λοιπόν ότι η διευκρίνηση αυτή ήταν χρήσιμη. Έχω πει ότι δεν, ήταν, δεν θα ήταν σκόπιμο να περάσουμε αυτή την περίοδο του ενός μηνός αλλά τώρα πάντως η διευκρίνηση έγινε. Ο κύριος Λάγκεν. Ε, ευχαριστώ. Ε, συζητούσα τώρα εδώ με την γειτόνισά μου και στη διάρκεια της τελευταίας σας φράσης. Σήμερα το πρωί, επανέρχομαι σε μια συζήτηση που κάναμε σήμερα για, την, για τα παράγωγα και για την ευρωπαϊκή ε, ασπίδα διάσωσης. Και εδώ τίθεται το θέμα της πρόσβασης σε χρήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αφενός, τι γίνεται με τα κέντρα συμψηφισμού, αν θα πρέπει να έχουν δηλαδή άδεια τραπεζικών δραστηριοτήτων ή να έχουν πρόσβαση σε χρήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και προκειμένου, εάν για το Ταμείο Διάσωσης του Ευρώ, άλλωστε έχετε αγοράσει και σε ύψος δισεκατομμυρίων κρατικά ομόλογα και αυτό, γι' αυτό έχετε επικριθεί κιόλα. και αν μέσα στα πλαίσια αυτού του Ταμείου Διάσωσης που μπαίνει τώρα στην φάση των δοκιμασιών, των τεστ και βλέπω να μην υπάρχει τέλο μετά από την Ελλάδα και την Ιρλανδία. Αν σύμφωνα με το άθρο 125 το οποίο ΆΘΟ απαγορεύει την αγορά κρατικών χρεών και ευρωομολογών κατά τη γνώμη μου αν λοιπόν κατά την άποψη σας υπάρχει μια δυνατότητα αναχρηματοδότησης του μηχανισμού διάσωσης μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν βλέπετε δηλαδή κάποια δυνατότητα το Ταμείο αυτό να μπορεί να χρησιμοποιήσει πόρους της ε, Κεντρικής Τράπεζας. Και το γεγονός ότι η Fed έχει επιλέξει διαφορετική ε, λύση γιατί μπορεί και αυτό να οδηγήσει σε κίνδυνο πληθωρισμού. Δηλαδή τώρα, πώς βλέπετε αφενός τα κέντρα συμψηφισμού στον τομέα των παραγόγων και το ενδεχόμενο το Δαμείο Διάσωσης να έχει πρόσβαση σε χρήματα της Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ, είναι εξαιρετικά σημαντικό το ερώτημά σας. Μάλλον ερωτήματα γιατί νομίζω ότι θέσατε, θίξατε πολλά θέματα. Αφενός τα κέντρα συμψηφού, τα clearing houses και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται με τη ρευστότητα της κεντρικής τράπεζας ή δεν συνδέονται. Είναι αυτούσιο το ερώτημα αυτό. Και πρέπει να ενταχθεί μέσα σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο γιατί πρέπει να εφαρμόζουμε τους ίδιους κανόνες σχετικά με τα clearing house στο παγκόσμιο επίπεδο. και αυτό συζητείται και στις κεντρικές τράπεζες των ανεπτυγμένων αλλά και των αναπτυσσομένων οικονομιών. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα καθεαυτό, ξεχωριστό. Και έχουμε τώρα και το ερώτημά σας, αν κατανοώ καλά, σχετικά με το πρόγραμμά μας αγοράς ομολόγων και είναι ένα από τα μη στάνταρτ μέτρα που αποφασίσαμε δεν έχω κανένα άλλο σχόλιο. Είναι απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών και η απόφαση αυτή λήφθηκε διότι θεωρήσαμε ότι οι διάβλοι μεταφοράς της νομισματικής πολιτικής παρεμποδίζονταν, παρακολύονταν στην προσπάθεια ε, να ε, αποκαταστήσουμε τους διάβλους αυτούς. Γνωρίζετε ότι δεν αλλά αλλάζουμε τίποτε διότι αφαιρούμε την ρευστότητα η οποία έχει διατεθεί μέσω του προγράμματος αυτού. Σήμερα το πρωί αποσύραμε πάλι την ρευστότητα η οποία είχε διοχετευτεί και αυτό το κάνουμε κάθε εβδομάδα. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί τώρα για το μέλλον. Είναι απολύτως απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών. Αλλά το πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται. Τώρα με ρωτάτε εάν θα είμαστε εμείς σε θέση να αναχρηματοδοτήσουμε το Ταμείο Διάσωσης. Το Ταμείο αυτό είναι πλήρως λειτουργικό, όπως γνωρίζετε. Εγκρίθηκε τον Μάιο και λειτουργεί για πρώτη φορά τώρα, διότι στην περίπτωση της Ελλάδος δεν ήταν αυτό το Ταμείο, το EFSF, ήταν με ε, ειδικά δάνεια, με ad hoc δάνεια. Δεν χρηματοδοτούμε εμείς οι ίδιοι το EFSF, που είναι ο μηχανισμός που είναι στα χέρια των κυβερνήσεων. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση σας, κύριε. Κύριε Πρόεδρε. Είπατε ότι η πολιτική ουσιαστικά είναι νομισματική, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Οικονομική Τράπεζα. Στις Ηνωμένε Πολιτείε ο κύριος στόχος είναι ο πληθωρισμός και η χαραγώγησή του. Η οικονομική πολιτική πολιτική ε, στην Ευρώπη πράγμα που δεν συμβαίνει στην Αμερική ε, επαφίεται στις κυβερνήσεις η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν φαίνεται να έχει διαφορετική και ε, αρμοδιότητες από ό,τι ισχύει στη, για τη ΦΕΔ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς πού βλέπετε τώρα, πώς βλέπετε τώρα να δρά και τι περιμένετε να κάνει στην πεδίο της οικονομικής πολιτικής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, ε, ε, έχει ακουστεί ότι δεν πρέπει ο μηχανισμός διάσωσης να είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο οποίο θα κολλήσουμε, θα κρεμάσουμε όλα τα δεινά που υπάρχουν και θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Τι γνώμη έχετε εδώ. Εδώ, απάντηση, εδώ πρόκειται για ένα θέμα διακυβέρνησης το οποίο αφορά στο πολύ μακροπρόθεσμο μέλλον της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη υπάρχουν 17 μέλη. Εσείς μιλάτε για μια Ευρωζώνη των 27, έτσι. Είναι λοιπόν πολύ μακροπρόθεσμο το όνειρό σας αυτό και η ιστορία της διακυβέρνησης που συζητιέται τώρα είναι πώς θα κάνουμε τη διακυβέρνηση όταν θα έχουμε 27 χώρες στο ευρώ, 330 εκατομμύρια κόσμο. Όμως, και όμως θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα μόνιμο το οποίο εάν και εφόσον δεν λειτουργεί καλά το σύστημα εποπτείας θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί. Η πιθανότητα μεμονωμένων χωρών και οικονομιών να μη λειτουργούν σωστά να μην ακολουθούν τους κανόνες και συγχρόνως να έχουμε και τους επίτροπους που δεν εποπτεύουν σωστά. Αυτή, η πιθανότητα να σημαίνουν και αυτά τα δυο και να οδηγηθούμε σε μια τελείως χαλαρή αν θέλετε διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μικρή Και αυτό το σενάριο δηλαδή προσπαθείτε να μου πείτε να σχολιάσω της ε, υπερβολικής χαλαρής αντιμετώπισης και από τους μεν και από τους δε. Όμως αυτό σας λέω είναι μάλλον απίθανο. Σε τελευταία ανάλυση Βεβαίως ξέρουμε ότι η κρίση ισχύει για όλους και όλες οι οικονομίες οι αναπτυγμένες αυτή τη στιγμή αναζητούν λύσεις και μέτρα για να διορθώσουν τα πράγματα να γίνει καλύτερη διαχείριση των οικονομικών πολιτικών και να μην επανέλθουμε γίνουν τα ίδια λάθη που μας οδήγησαν εδώ υπάρχει αυτή η πίεση λοιπόν και βεβαίως ευτυχώς τώρα μπήκαμε μέσα σε μια κρίση αλλά δεν είναι ίδια κρίση όπως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ε. Πρόεδρος Νομίζω ότι δεν λειτουργούμε σωστά από άποψη χρόνου. Η Ελίζα Φερέρα είναι η επόμενη ομιλήτρια. Θα είστε λίγο σύντομοι. Ε? Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Το βασικό μου ερώτημα σχετίζεται με τον ε, μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Λειτουργεί αλλά δεν φτάνει στους απότερους στόχους. Ε, δηλαδή μολύνθηκαν και άλλες χώρες, αυτό δεν αποφεύχθηκε και φαίνεται ότι δεν έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών. Θα ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο της ΕΚΤ πώς θα το αντιμετωπίσει, διότι η ΕΚΤ είναι σταθεροποιητικός παράγων, αλλά ποια θεωρείτε ότι είναι τα αίτια του ότι ο μηχανισμός αυτός δεν εκπλήρωσε τους απότερους στόχους του. Υπάρχει ένα ε, θέμα διακυβέρνησης και ένα ζήτημα διακρατικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, που δεν είναι το κουτί της Πανδώρας. Θα ήθελα να μας πείτε πώς σκέφτεστε σε σχέση με το μακροχρόνιο χρέος ορισμένων χωρών. Μπορούν να διαχειριστούν ένα πλεόνασμα το οποίο να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την αποπληρωμή αυτού του χρέους. Πιστεύετε ότι η Ευρωζώνη μπορεί να ανταποκριθεί, διότι έχουμε να κάνουμε με χώρες που έχουν διαφορετική παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Νομίζω ότι το κύριο θέμα, ως συνήθως, είναι η σχετική ανταγωνιστικότητα μεταξύ των διαφόρων χωρών. Αυτή θα πρέπει να, την κατάσταση θα πρέπει να την παρακολουθούμε. Έχω πει επανειλημμένος στις ε, συναντήσεις και τις που οργανώσατε ότι είμαστε σε μια ενιαία περιοχή με μια ενιαία αγορά με ένα ενιαίο νόμισμα όπου υπάρχει όμως σταθερότητα τιμών γύρω στο 2% τα τελευταία χρόνια και όπου η σταθερότητα αυτή θα παραμείνει στην επόμενη δεκαετία. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί που παίρνουν αποφάσεις, κοινοβούλια, ε, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, γιατί αυτό είναι θεμελιώδες. Είμαστε στην ίδια ενιαία περιοχή και οικονομία και έχουμε και ένα benchmark το οποίο είναι η ονομαστική εξέλιξη, ανάπτυξη. Για τη σταθερότητα τιμών λοιπόν 1,97, 2% περίπου. Όλοι εδώ μέσα αυτό το πλαίσιο θα πρέπει λοιπόν να ανταγωνίζονται όλοι. Όσον αφορά την παραγωγικότητα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα παραγωγικότητας. Αλλά ανάλογα με το επίπεδο της παραγωγικότητας προσαρμόζει κανείς τις αμοιβέ και το κόστος του ώστε να μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστικός. Αυτό το κάνουν όλες οι οικονομίες του κόσμου. Αυτό πρέπει να γίνει, να γίνεται όταν κανείς ανήκει σε μια ενιαία περιοχή ενιαίου νομίσματος. Εκείνο που μετρά λοιπόν είναι το μοναδιαίο κόστος εργασίας. Ε? Αυτό μετράει για τον ανταγωνισμό, ε? για την ανταγωνιστικότητα. Πρόεδρος, θα πρέπει να περιοριστούμε στα τέσσερα λεπτά ένα θέμα, ε? ενάμιση και δυόμιση ε, λεπτά. Το Κοινοβούλιο προσπαθεί να αναλάβει τις ευθύνες του. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι κάνανε οι χώρες της Ευρωζώνης δεν χρειάζεται να μας πείσετε μας. Πείστε την αγορά, τις αγορές. Γιατί λέτε ότι φτάσαμε στα σωστά διδάγματα μετά από την κρίση του πρώτου ή δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Έτσι μας είπατε. Ε, και γνωρίζουμε ότι υπάρχει η ευρωπαϊκή πολιτική αλλά και οι εθνικές πολιτικές γιατί έχουμε να κάνουμε με μία ονέ από τη μία πλευρά αλλά έχουμε να κάνουμε και εθνικές πολιτικές. Έχουμε διαφορετικές φορολογικές πολιτικές, ε, πολιτικές κόστους της εργασίας, άρα δεν υπάρχει ε, ίση πρόσβαση. Τι πρέπει να κάνουμε, να εποπτεύσουμε τις διαφορές, ίσως θα ήταν καλύτερα από την ενοποίηση. Δεύτερον, με εκπλήσει το εξής. Το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή έχει την τάση να μειώνει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 10 Ιουνίου η ΕΚΤ είχε προβεί σε μία ανακοίνωση για, για το πώς θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε σε αυτό το πακέτο. Και υπήρχε ένας ε, κανονισμός που αφορούσε την εξυγίανση και την αντιμετώπιση της κρίσης. Και τώρα μας λέτε όχι, αυτό το θέμα αφορά το Συμβούλιο. Δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να επανεισαγάγουμε και το θέμα των ε, κρατικών, του κρατικού χρέους, του δημόσιου χρέους και όπως είπε και ο κύριος Μαργκάγιο να δούμε πώς μπορούμε να εξηγιάνουμε τον τομέα των τραπεζών. Ναι, Σάρων, αλλά θα ήταν σκόπιμο, μια και έχουμε τον κύριο Τρισέ μαζί μας, εδώ μεταξύ μας να αδράξουμε την ευκαιρία. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για εξυγίαση των τραπεζών, κάτι το οποίο ποτέ δεν αποφασίστηκε και το οποίο στοιχίζει ακόμα περισσότερο στους φορολογούμενους. Ως προς το πρώτο σας σχόλιο, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα. Και εμείς θεωρούμε ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι ανεπαρκής και ξέρουμε ότι το Συμβούλιο είχε καθυστερήσει να απαντήσει στην πρόταση της Επιτροπής. Εσείς είσαστε η... ο νομοθέτης και θα σας απασχολήσει το ζήτημα. Εγώ μίλησα για ιονή ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο εάν υπάρχει ενισχυμένη εποπτεία σε σχέση με την παρούσα διάχυτη κατάσταση, η οποία δεν αντικατοπτρίζει πλήρως αυτά τα δεδομένα. Εδώ χρειαζόμαστε ε, μία ε, ιονή δημοσιονομική πολιτική ομοσπονδιακού χαρακτήρα. Ως προς την επίλυση κρίσεων, και εδώ σας μιλώ από καρδιάς, Είχαμε τόσο μεγάλες δυσκολίες για να αποσαφηνίσουμε το όλο πλαίσιο, ώστε δεν θέλω να ανοίξω για άλλη μια φορά το κουτί της Πανδώρας. Βεβαίως ε, εξαρτώμε από την κρίση του Κοινοβουλίου και τη θέλησή του. Θα πρέπει να είμαστε συνετοί, έχει αποσαφινιστεί η κατάσταση και αυτό το στοιχείο είναι ύψης της σημασίας ως προς την, ε, τις τράπεζες. Εσείς λάβατε πολύ σημαντικές αποφάσεις για μια γενικότερη αναθεώρηση. Βεβαίως απέχει από μια ιδεατή κατάσταση που θα επιθυμούσαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, έχουμε τις εθνικές εποπτικές αρχές, έχουμε τον οδικό χάρτη για την ε, προληπτική εποπτεία, ας τα θέσουμε αυτά σε εφαρμογή. Το λόγο έχει ο κύριος Ντάκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις για το Βέλγιο γιατί υπάρχει μεγάλη πολιτική αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή στο Βέλγιο υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία ασχολείται με την καθημερινότητα αν θέλετε με τα, την καθημερινή διακυβέρνηση της χώρας ε, αλλά η κατάσταση είναι τέτοια που υπάρχουν ερωτηματικά για το κατά πόσο θα συνεχίσει να υφίσταται το Βέλγιο ως κράτος. Εγώ δεν έχω άποψη. Πραγματικά ε, εγώ ρωτώ τώρα για το τι γίνεται σε σχέση με το Βέλγιο τι, πώς συνδέεται την πολιτική αβεβαιότητα και μη σταθερότητα στο Βέλγιο και το ερωτηματικό αν θέλετε σχετικά με την ύπαρξή της και την άλλη μεριά την αντιμετώπιση των αγορών όπου βλέπουμε επιτόκια 12,5% στη Γερμανία και 3,5% στο Βέλγιο απάντηση. Παρατηρώ τι γίνεται στις διάφορες χώρες. Πρέπει να το παρατηρήσουμε. Και πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας. Δεν ε, νομίζω ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της πολιτικής αβεβαιότητας στο Βέλιο και της ε, στάσης των αγορών. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Από εκεί και πέρα σε πολιτικό επίπεδο μπορεί να υπάρχει πρόβλημα και εσείς πολιτικοί αυτά τα ξέρετε ακόμη περισσότερο από μένα ε, πρέπει να ενημερώνεται ο πολίτης να ε, βλέπει πώς ε, λειτουργεί ο κόσμος γύρω του, να συνειδητοποιεί γιατί και πώς. Αυτό είναι πιο σημαντικό για το Βέλγιο αυτή τη στιγμή από ότι ίσως για άλλες χώρες. Γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ υψηλό ε, χρέος. Πρέπει λοιπόν να εξηγιάνουμε την κατάσταση το 2008 και το 2009 το 2009 με την Ελλάδα και το 2010 με την Ιρλανδία έπρεπε να προσφύγουμε στο τραπεζικό τομέα. Βεβαίως οι δανειοδότες και οι δανειολήπτες φέρουν, φέρουν ευθύνη. Και τέλος, ποιος καταβάλει το αντίτιμο, οι φορολογούμενοι και ιδιαίτερα οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση εξαιτίας των αγορών. Θεωρείται ότι θα πρέπει να αρκεστούμε σε παρόμοιες λύσεις. Εσείς μα λέτε ότι η οικονομία βαίνει καλώς και τα 27 κράτη-μέλη έλαβαν μέτρα λιτότητας. Αυτό δεν ισχύει γιατί μερικές χώρες δεν έχουν λάβει μέτρα λιτότητας. Και στις χώρες όπου υπάρχει αυστηρή λιτότητα δεν μπορούμε να πούμε ότι η οικονομία βαίνει καλώς. Αυτά τα μέτρα δεν είναι αντιπαραγωγικά και δεν οδηγούν στον αποπληθωρισμό. Μιλάτε για maximum boldness, ότι δηλαδή θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα τολμηροί, ιδιαίτερα θαραλέοι για να εξημερώσουμε τις κυβερνήσεις. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να εξημερώσουμε τους άλλους οικονομικούς φορείς που έδρασαν ανεύθυνα διότι αυτό αφορά τον, τραπεζο, τραπεζο, τον χρηματοοικονομικό τομέα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και η ΕΚΤ θα πρέπει να δράσει θαραλέα για να πατάξει τους κερδοσκόπους των τραπεζών. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω από τις τελευταίες σας ερωτήσεις. Οι οικονομίες δεν βαίνουν καλώς, μερικές τουλάχιστον. Μερικές τα πάνε υπερβολικά καλά. Σε μερικές περιπτώσεις ή πήγαιναν υπερβολικά καλά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την αντίστροφη κατάσταση από δημιουργίας ευρώ. Δηλαδή έχουμε οι οικονομίες που πάνε πολύ καλά τώρα, αλλά που είχαν να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες αποκατάστασης του ανταγωνισμού, ως όσον αφορά τον ανταγωνισμό τους, και άλλες οικονομίες που δεν βαίνουν καλώς τώρα, που τα πήγαιναν καλά στο παρελθόν. Ξέρετε πού αναφέρομαι. Αναφέρομαι και στις ΗΠΑ. Υπάρχει δηλαδή μια αντιστάθμιση ε, μεταξύ εκείνων που πήγαιναν καλά στο παρελθόν και όχι τώρα και το αντίστροφο. Εκείνων που πήγαιναν καλά στο παρελθόν και όχι πλέον. Εκεί θα πρέπει να γίνει μια ανασύνταξη. Δεν θέλω να δημιουργήσω την εντύπωση ότι είμαι συγκαταβατικός. Ε, γνωρίζουμε δύσκολους καιρούς. Δεν μπορούμε να είμαστε συγκαταβατικοί αλλά στα πλαίσια της ε, πραγματικής οικονομίας δεν μπορώ παρά να πω το εξής. Από την ε, στιγμή της επαναφοράς της ανάπτυξης, μετά από αυτή την ύφεση που ήταν η πιο σημαντική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ε, μας εξέπληξε η κατάσταση σε σχέση με τις προβλέψεις, δηλαδή είναι λίγο καλύτερη από την προβλεπόμενη. Μήνα προς μήνα το βλέπουμε αυτό. Θα εκδώσουμε τις επόμενες προβλέψεις μας σε δύο μέρες, αλλά μέχρι ε, του παρόντος έτσι είχε η κατάσταση. Ως προς το άλλο σχόλιο σας, μάλλον ως προς το, τη συνολική σας παρατήρηση, ότι ζητάμε μερικοί να καταβάλουν προσπάθειες ενώ όχι άλλοι. Εδώ θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Δεν πρέπει να υπάρχουν αμφισημίες. Θα πρέπει οι πιστωτές να πληρώνουν. Αυτό τι σημαίνει. Ε, ότι εκείνοι που έδειξαν εμπιστοσύνη στην αγορά χάνουν χρήματα και εκείνοι που δεν συμβάλλουν στην αγορά θα πρέπει να κερδίσουν. Όλα είναι πιο περίπλοκα από όσο φαίνονται. Δεν πρέπει να απλουστεύουμε τα πράγματα. Οι σημερινές αγορές ε, έχουν να κάνουν με εκείνους που συνεισφέρουν πολύ και σε εκείνους που συνεισφέρουν πολύ λίγο. Γι' αυτό θα πρέπει να προβούμε στις ανάλογες αντισταθμίσεις για να υπάρχει εξισορρόπηση. Γι' αυτό θα πρέπει να ισχύσουν οι κανόνες που ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Είτε ε, αναλύουμε την κατάσταση όπως κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που λέει ότι η κατάσταση είναι βιώσιμη τότε υπάρχει υποστήριξη και από τους Ευρωπαίους, εάν το επιθυμούν. Και υπάρχει και η άλλη περίπτωση που δεν θεωρούμε πιθανή και θα σας μιλήσω για το τι είπαν οι κυβερνήσεις. Στην απίθανη περίπτωση όπου μια χώρα είναι αφαιρέγγια, in the unexpected event. Θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια λοιπόν, γιατί δεν μπορούμε να αποστέλουμε μηνύματα που είναι αντιφατικά. Γι' αυτό θεωρώ ότι η αποσαφήνιση ήταν πολύ σημαντική που έγινε από τις κυβερνήσεις. Ορίστε Φίλιπ, ζητήσατε πάθος στη συζήτηση. Να και το πάθος. Νίκολας. Νίκολας, συγγνώμη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που είστε άλλη μια φορά κοντά μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε αυτές τις στιγμές στη συνεδρίασή μας. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να κάνω μια επίκαιρη ερώτηση που μας απασχολεί στην Ελλάδα αυτές τις ώρες. Μετά την προκτεσινή εκτίμηση του ΕΚΟΦΗΝ στις 28 Νοεμβρίου ότι θα εξετάσει την πιθανότητα επέκτασης της προθεσμίας αποπληρωμής του δανείου που έλαβε η Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις χώρες τη Ευρωζώνης, μια τέτοια επέκταση θεωρείται δεδομένη στα ελληνικά πολιτικά πράγματα μέχρι το 2021-2024. Όμως το πρόβλημα που μας απασχολεί, απασχολεί την ελληνική κοινωνία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχω τις περισσότερες εφημερίδες μπροστά μου, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξή. Μια τέτοια επέκταση της αποπληρωμής σημαίνει ότι θα έχουμε επέκταση και της λιτότητας που επέφερε το μνημόνιο που συνήψει η Ελλάδα με τις Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν λάβετε υπόψη, κύριε Πρόεδρε, ότι ορισμένοι δείκτες κατά την πρόβλεψη της Κομισιόν δεν θα πάνε καλά, όπως το δημόσιο χρέος, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πράγματι επιμήκυση του μνημονίου. Ή να το διατυπώσω διαφορετικά. Θεωρείτε πιθανόν ότι θα υπάρξει ένα τέτοιο μνημόνιο λιτότητας και μετά το 2013 για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Nous avons nos responsabilités. We have our... Φέρουμε ευθύνη, μεγάλες ευθύνες όπως γνωρίζετε. Όλα τα ερωτήματα που θέσατε είναι ερωτήματα για τις κυβερνήσεις, δεν είναι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τράπεζας. Δεν θα ήθελα λοιπόν να πω κάτι τι, το οποίο να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, διότι ακούγονται πολλές φωνές, πολλαπλές φωνές και ο καθένας μιλάει για, λέει τα δικά του. τα ερωτήματα λοιπόν είναι ερωτήματα για τις κυβερνήσεις, για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και για την Κομισιόν ίσως που επιβλέπει. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού, της ελληνικής οικονομίας να επανέλθει μονίμως σε μία νορμάλ λειτουργία της αγοράς. Αυτό η λιτότητα, η λιτότητα τι σημαίνει. Όταν είχαμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα συμπεριφοράς μη νορμάλ, ε, πρέπει να επανέλθουμε σε μια κατάσταση νορμάλ. Δεν είναι ακριβώς λιτότητα λοιπόν. Back to normal. Να επανέλθουμε στις κανονι... στην κανονική λειτουργία της αγοράς. Με... Ε, σοβαρές πολιτικές μακρό, μη, μακροπρόθεσμες. Thank you, Chair. In an interview... Μάρτα σε μια συνέντευξη στο Le Progrès που δώσατε λίγο πριν, είπατε ότι η έννοια των κυρίαρχων κρατών δεν βρίσκει πραγματικό αντίκρισμα σήμερα στον πραγματικό κόσμο αυτή η φιλοσοφία σας επηρεάζει στην στάση σας ως Προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας και αν ναι μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το ε, κυρίαρχο εθνικό κράτος είναι και σωστή ε, δομή ο Πρόεδρος. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Είπα ότι έχουμε δημιουργήσει νέες οντότητες οι οποίες είναι σημαντικές είτε παγκόσμια είτε στο επίπεδο της Υπήρου. Γνωρίζουμε τώρα ότι ένα γεγονός στη, για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να θέσει σε εκείνες τις διαδικασίες που επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο και ότι πρέπει να ε, φτιάξουμε επίπεδα διακυβέρνησης στο παγκόσμιο επίπεδο που θα συμβαδίζουν με την ύπαρξη αυτής της νέας οντότητας που είναι η παγκόσμια οικονομία και τα παγκόσμια δημοσιονομικά και πρέπει να είναι και συντονισμένα με αυτά που εξακολουθούν να παραμένουν τα θεμέλια των κυρίαρχων κρατών, δηλαδή, όπως έλεγα, η συνθήκη της Βεσφαλίας που δημιούργησε στην Ευρώπη αυτή την έννοια του κυρίαρχου κράτους. Είναι λοιπόν αληθές το ίδιο και για την Ευρώπη, που είναι και πολύ πιο φιλόδοξη για το παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε όμως μια ενιαία ευρωπαϊκή οικονομία και μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και αυτό ήταν και ε, το φιλόδοξο σχέδιο των ιδρυτών πατέρων και έχουμε όπως είπα μια ενιαία αγορά με ένα κοινό νόμισμα. Και είναι αυτός ο συνδυασμός νέων οντοτήτων που είναι πάρα πάρα πολύ ε, σημαντικές τώρα πλέον και αυτή η βεσφαλική εντός εισαγωγικών έννοια της ε, κυριαρχίας του κράτους. Εσείς όμως εδώ είστε η ενσωμάτωση, είστε η προσωποποίηση ε, αυτής της έννοιας της συνεργασίας των βεστιφαλικών κυριαρχών κρατών και της ανάγκης να ε, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες οντότητες 500 εκατομμύρια άνθρωποι και 27 χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Hans Peter Martin. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αποφύσει το αξιώματο σας κύριε Πρόεδρε. Λέτε ορισμένα πράγματα τα οποία ίσως έχουν διαφορετικό νόημα. Θυμάμαι πριν από ένα χρόνο πώς ήταν τα πράγματα με την Ελλάδα. Σήμερα θα αναφερθώ στην Ισπανία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε, γνωρίζουμε ότι έχει σχετικά μικρό κρατικό ε, χρέος ωστόσο έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα επίπεδα του δανεισμού. Και αυτά που συμβαίνουν ε, γενικά στη χώρα αυτή δεν φαίνεται να είναι ε, τρομακτικά, αλλά φαίνεται άλλοι να γνωρίζουν περισσότερα πράγματα από εμείς. Φαίνεται να υπάρχει μια κρεμότητα 100 δισεκατομμυρίων ε, ευρώ και τα πράγματα ε, φαίνεται να ρυθμίζονται πολύ διαφορετικά στην Ισπανία από ό,τι ε, σε κεντροευρωπαϊκές χώρες. Ίσως λοιπόν τα πράγματα να αρχίσουν να εμφανίζονται σε 5 ή 10 χρόνια εκεί. Ερώτηση, έχετε μια ρεαλιστική ε, αξιολόγηση της κατάστασης των ε, οικοδομικών πιστώσεων, των πιστώσεων δηλαδή για την οικοδομή στην Ισπανία. Και μπορείτε να φανταστείτε εάν μία από τις μεγάλες ενοποιημένες τράπεζες, Σανταντέρ ή κάποια άλλη, πτωχεύσει, ε, ποιες μπορείς να είναι επιπτώσεις. Θα ήθελα να θυμηθούμε όλοι ότι εκ της συνθήκης καλούμεθα να εξασφαλίσουμε τη νομική σταθερότητα 16 χωρών και 300 περίπου εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό είναι η εντολή μας. Αυτό που κάναμε επί 12 χρόνια με 1,97% ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού. Η σταθερότητα των τιμών εξασφαλίζεται καλύτερα στην ζώνη ευρώ σε πλήρη συμμόρφωση με τη συνθήκη σε πλήρη συμμόρφωση με αυτά που μας ζητήσατε και πολύ καλύτερα από παλαιότερα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και για τα επόμενα δέκα χρόνια θα εξασφαλίσουμε την ίδια νομισματική σταθερότητα. Αυτή είναι η εντολή μας τα ερωτήματά σα είναι απολύτως εκτός της εντολή μα, απολύτως εκτός των ευθυνών μας και αρμοδιοτήτων μας και θα πρέπει να απευθύνονται σε άλλου φορεί. Το λέω καθαρά. Είπα ο ίδιο ότι δεν θα πρέπει να μιλούμε από εδώ και από εκεί. Χρειάζεται κάποια πειθαρχία στα λόγια. Είναι απόλυτα σημαντική λοιπόν αυτή. Δεν είμαι υπεύθυνο τη οποιασδήποτε χώρα χύψη δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εποπτεία των διαφόρων χωρών. Βρισκόμαστε σε επαφή, σε σύνδεση με τις υπεύθυνες αρχές, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφενός και το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών από την άλλη. Είπαμε πάντοτε σε όλες τις χώρες ότι προσοχή θα πρέπει να κάνετε την πιο σόφρονα και λογική διαχείριση. Αυτό μας ακούσατε να λέμε διαρκώς. Έχοντας πει αυτό θα είπα ακόμη ότι ένας αριθμός παρατηρητών πιθανώς υποτίμησαν την ε, υγεία της Ευρωζώνης στο σύνολό της, καθώς και πολλών χωρών, και ίσως είναι ένας συνδυασμός. Πώς να το πω. Ίσως μιας επικοινωνιακής αμφισημίας αυτό που χρειάζεται είναι να επανέλθουμε ε, στην πιο ξεκάθαρη και ακριβή επικοινωνία. Μίλησα προηγουμένως για χρήσιμες διευκρινήσεις. Δεν θεωρώ διόλου ότι η υπόθεση εργασίας που προβάλλεται για τις ε, ισπανικές τράπεζες είναι καθόλου ρεαλιστική. Obrigado. Muito obrigado, σας ευχαριστώ για την ε, πολύ ζωηρή σας παρέμβαση. Στην, πρόταση, στην πρώτη σας ε, παρέμβαση μιλήσατε για το πακέτο της Επιτροπής για την ε, χρηστή διακυβέρνηση και μας είπατε ότι η ΕΚΤ είχε αμφιβολίες ως προς ορισμένες προτάσεις που θα οδηγούσαν σε ε, διακρίσεις, ιδιαίτερα στον ε, έλεγχο του χρέους εξάντε. Και γι' αυτό ακριβώς θα έπρεπε να δούμε ποιες είναι οι έκτακτες οικονομικές συνθήκες. Ε, θα θέλατε να διαγραφεί αυτή η μνήα ή προβάλλεται μια εναλλακτική διατύπωση. Ως προς το θέμα του ανταγωνισμού τώρα. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα, την Πορτογαλία, που έχει ένα πολύ αυστηρό εργατικό δίκαιο. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ευελιξία στον τομέα αυτό του εργατικού δικαίου και να ισχύσουν ευρύτεροι κανόνες που να οδηγήσουν και σε υψηλότερο ανταγωνισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ ήμουν νομίζω σαφής. Είπα ότι θέλουμε να ενισχυθεί ακόμη και το κείμενο της Κομισιόν για τη διακυβέρνηση και προσπάθησα να δώσω και παραδείγματα για το που θα πρέπει να ενισχυθεί, να γίνει πιο έντονο το κείμενο της Κομισιόν. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες βεβαίως γιατί είναι ρευστό, ε, εξελισσόμενο το κείμενο οπότε ε, δεν θέλω να κάνω σχόλια. Αλλά είναι νομίζω απολύτως σαφές ότι σε όλες τις χώρες δίχως εξαίρεση ακόμη και σε εκείνες που ε, τα πάνε καλά σήμερα ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εξέλιξη, την οικονομία μελλοντικά και στην Πορτογαλία. Λέω λοιπόν ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές στην Πορτογαλία ακόμη και στην αγορά εργασίας θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην Πορτογαλία να ξεπεράσει τα προβλήματά της πιο καλά πραγματικές διαρθρωτικές αλλαγές είναι πολύ σημαντικές για όλους πέραν των ε, σταθερών, στέρεων και αυστηρών πολιτικών για το μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η απάντηση λοιπόν είναι ναι. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που αναγνωρίζετε πλήρως το, τον νομοθετικό ρόλο του Κοινοβουλίου στη, ε, στο θέμα της διακυβέρνησης. Είναι καινούριο ο ρόλος η αρμοδιότητα αυτή για το, για το Κοινοβούλιο. Έχω δύο ερωτήσεις να σας κάνω κύριε Τρισέ. Πρώτη ερώτηση. Είναι προφανές ότι υπάρχει σημαντική αναταραχή στις αγορές ακόμη και δεν είμαι πεπισμένη ότι η Ιρλανδία είναι η τελευταία χώρα που, την οποία πρέπει να διασώσουμε. Είναι έτσι. Δεύτερο, πιστεύετε ότι το πακέτο νομοθετικών προτάσεων μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα και υπάρχει σχέση μεταξύ με, με το νέο στα, μηχανισμό τα της Ελλάδας θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε ποια είναι η σχέση του μηχανισμού αυτού με το, με τη, το νομοθετικό πακέτο μήπως θα πρέπει να περιμένουμε πριν να πάρουμε οριστική απόφαση Τρισέ. Κατάλαβα τι εννοείτε. Και απλώς θα σας δώσω τη δική μου άποψη. Έτσι όπως το αισθάνομαι εγώ. Βεβαίως, όπως είπα, αγαπάμε τους δημοκρατικούς μας θεσμούς και υποστηρίζουμε τη δημοκρατία με κάθε τρόπο. Η αίσθησή μου είναι ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη αυτή τη στιγμή ε, γιατί επειδή υπάρχει αβεβαιότητα δόθηκαν σαφείς εξηγήσει. δεν προτείνω να ξανανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας αυτή τη στιγμή αλλά καταλαβαίνω που λέτε τι, τι υπονοείτε με αυτό που λέτε. Τώρα, για την ανίσχυση του κειμένου και στο φορολογικό κομμάτι, το δημοσιονομικό και στο κομμάτι της εποπτείας, αν προχωρήσει κανείς όσο το δυνατόν γίνεται προς αυτήν την ιονή ομοσπονδιακή κατάσταση Ά, ένα είδος Βεσφαλίας κυρίαρχα κράτη γύρω από μια κεντρική εξουσία ε, αν μπορέσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε ως το δυνατόν περισσότερο προς αυτή την ιωνία ομοσπονδιακή κατάσταση, το καλύτερο, αλλά εσείς είστε ο νομοθέτης, δεν είναι δικό μου θέμα. Βέβαια αυτή τη στιγμή μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί είναι καινούργια ιδέα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε αν τα αποφασίσετε. <laughs> Δεν ανησυχώ. Right, Burkhard, it's your go now. Uh, ich habe... Κύριε Πρόεδρε, δύο σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πώς βλέπει το μελλοντικό της ρόλο στον χαρισμό κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι ε, τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν τα πάει άσχημα αλλά τώρα καλείται να αναλάβει και καινούργια ε, καθήκοντα έχει αγοράσει ε, τεράστια ε, ποσά από τις διάφορες χώρες πώς βλέπετε το μελλοντικό της ρόλο λοιπόν δεύτερο ερώτημα ευρωομόλογα η ιδέα αυτή όλο και πιο επίκαιρη γίνεται και πάλι Βεβαίω υπάρχουν αυτοί που είναι υπέρ, υπάρχουν αυτοί που είναι κατά. Σε ορισμένα κράτη μάλλον θεωρείται και αντισυνταγματικό κάτι τέτοιο ακούστηκε ότι τα ευρωμόλογα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ε, χρηματοδότηση του 60% μοναχά των ε, χρεών των κρατών μελών. Τι να σας πω, ε, αν διαχωριστεί έτσι η αγορά, πιστεύετε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, ποια είναι η άποψή σας. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Όπως έχω πει, το θέμα δεν είναι... Ε, ε, ε, αυτό που κάνουμε με τις διάφορες χώρες είναι ότι αφαιρούμε και ξαναδίνουμε τη ρευστότητα αφαιρούμε τη ρευστότητα που δώσαμε κάθε εβδομάδα για να βοηθήσουμε λιγάκι τις αγορές όταν έχουμε μια οικονομία η οποία δεν λειτουργεί σωστά. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω αυτά που λέγονται από εδώ και από εκεί. Όπως ξέρετε, μέχρι τώρα δεν είμαστε εμείς που προωθήσαμε την ιδέα των ευρωομολόγων. Βεβαίως ποτέ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα, αλλά δεν θεωρήσαμε ότι υπήρχε ανάγκη για τα ευρωομόλογα. Οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα ακολουθούσαν άλλες άγουσες και η ιδέα αυτή του 60% ανεχρηματοδότηση μόνο του 60% δεν έχω καμία γνώμη. Δεν σχολιάνω από αυτό. Παρακαλώ. Oui, monsieur le Président. Κύριε Πρόεδρε, η κρίση καθιστά ε, σκόπιμη και απαραίτητη την παρέμβαση. Η ΕΚΤ δεν καταπολεμά μόνο τον πληθωρισμό και ο πρόεδρος της ΕΚΤ προβαίνει σε συστάσεις ως προς μία δημοσιονομική πολιτική, αν και δεν είναι υπεύθυνος για αυτή. Συστάσεις που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για νομισματικό πραγματισμό της ΕΚΤ έτσι ώστε να αποφύγουμε την κρίση της ρευστότητας, έτσι ώστε οι ιδιωτικές τράπεζες να αγοράσουν ένα μέρος του εθνικού χρέους και η ίδια η ΕΚΤ αγόρασε το δημόσιο χρέος του ελληνικού κράτους και το ίδιο έκανε και για περιφερειακές χώρες. Δύο ερωτήσεις λοιπόν θα ήθελα να υποβάλω. Εάν το θέμα του δημόσιου χρέους επεκταθεί στην Πορτογαλία, η ΕΚΤ θα αγοράσει ένα μέρος του χρέους της Ισπανίας ή της Πορτογαλίας, όπως κάνουν και οι ΙΠΑ γιατί είναι το πιο αποδοτικό μέσο για να αποσυμφορήσουμε τα επιτόκια στην αγορά ομολόγων. Επίσης, οι ισοτιμίες θα πρέπει να βοηθήσουν στην ισορροπία των νομισμάτων. Ένα ευρώ δηλαδή 1,17 δολάριο. Η ΕΚΤ θα παρέμβει εάν το Συμβούλιο της το ζητήσει και όπως επιβάλλει η συνθήκη της Λισαβόνας. Έτσι ώστε η ΕΚΤ όπως και η ΦΕΔ να παρέμβει άμεσα. Ποια είναι η άποψή σας? Sur la première question. Ως προς το πρώτο ερώτημα, θα ήθελα απλώς να σας πω ότι η απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών ήταν να ενταχθούμε σε αυτό το πρόγραμμα έτσι ώστε να συνεισφέρουμε για την καλύτερη λειτουργία του μηχανισμού νομισματικής πολιτικής. Έχουμε ένα εβδομαδιαίο δελτίο για τις παρεμβάσεις μας, τις χρηματοπιστωτικές παρεμβάσεις για να δούμε τι ρευστότητα βάζουμε στην αγορά με βάση αυτές τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Δεν έχω πρόθεση να πω τίποτα περισσότερο ως προς αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύουμε ότι εάν λάβουμε υπόψη το χρηματοοικονομικό περιβάλλον, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος παρέμβασης. Όσον αφορά τις ισοτιμίες, όπως είπα και πριν, έχουμε, αντιμετωπίσουμε δύο κύρια προβλήματα. Το ένα δεν είναι καινούριο. Αφορά την διακύμανση των μεγάλων νομισμάτων των αναπτυγμένων χωρών και αυτή τη στιγμή υπάρχει ελεύθερη διακύμανση, ελεύθερη διαμόρφωση, όπως γνωρίζετε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συνεχιστούν οι συζητήσεις στα πλαίσια αυτής της μικρής ομάδας αρχών, δηλαδή κεντρικών τραπεζών και κυβερνήσεων των νομισμάτων για να ορίσουμε τις ισοτιμίες μέσα στα πλαίσια αυτής της διακύμανσης των μετατρεπόμενων νομισμάτων. και αυτό έχουμε συμφωνήσει και στις διαβουλεύσεις με τους άλλους εταίρους, με την Ιαπωνία, της ΙΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Όσον αφορά τα νομίσματα των αναδυόμενων χωρών που έχουν μεγάλο πλεόνασμα, σας είπα ότι υπάρχει συνένεση και θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Ευχαριστώ. Ρόμπερτ. Κύριε Πρόεδρε, η ΕΚΤ επιτρέπει στις τράπεζες να επαναχρηματοδοτούνται με μια ισοτιμία που είναι στο ιστορικά χαμηλότερο, ε, χαμηλότερο, χαμηλότερη στάθμισή. Ε, στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Τι θα γίνει όμως από πλευράς αποταμιευτών διότι βλέπουμε ότι και στην περίπτωση δανειοδότησης η κατάσταση είναι απελπιστική. Η Κίνα δεν αγοράζει πια δολάρια από την αρχή του έτους, ε, αλλά δεν αγοράζει ούτε και ευρώ. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω αυτό που είπατε. Νομίζω ότι θα έπρεπε να θέσετε το ερώτημα στις κινέζικες αρχές. Όσον αφορά τις τράπεζες, θεωρούμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της οικονομίας αγοράς, της δικής μας οικονομίας αγοράς. Και δεν θα αποφανθώ επί αυτού που θα αποφασίσει το Συμβούλιο των Διοικητών στο μέλλον. Εν πάση περιπτώσει, τα επιτόκια μας συμβαδίζουν με μία αναγκαιότητα σταθερότητας τιμών. Για τις τραπεζές μας έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα εποπτείας των τραπεζών. Υπάρχουν και τα εθνικά εποπτικά συστήματα. Τώρα λειτουργεί αυτή η εποπτική αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η πολιτική θα εγγενιαστεί τον Ιανουάριο Υπάρχει και η οικονομία της αγοράς. Εσείς λέτε ότι οι τράπεζες κερδίζουν πολλά και αυτό δεν αντικατοπτρίζει τα χαμηλά επιτόκια. Κάποιος άλλος βουλευτής μίλησε για πιο δυσχερή κατάσταση την οποία αντιμετωπίσουμε ως προς τη δυνατότητα κέρδους, κερδοφορίας και ε, ίδιων πόρων. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολυσχηδή οικονομία της αγοράς και θα πρέπει ε, να ε, προωθήσουμε και να ενισχύσουμε αυτή την εποπτική διαδικασία και αρχή. Ο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, τις τελευταίες ημέρες η ρευστότητα ε, δυστυχώς έχει λήξει και πολλοί οι οικονομικοί φορείς μιλάνε για παρόμοια κατάσταση που γνωρίσαμε στην αγορά ομολόγων το 2007-2008. Ποια είναι η απόψή σας την ε, προηγούμενη εβδομάδα ο Επίτροπος Αλμούνια είπε ότι η Ισπανική κυβέρνηση θα πρέπει να αποσαφηνίσει την κατάσταση των αγορών σε σχέση με την αναθεώρηση ε, της, ε, της οικονομικής κατάστασης στην αγορά και την αναδιάρθρωση της κατάστασης. Απάντηση. Όπως ξέρετε δεν ε, σχολιάζω την λειτουργία της αγοράς σε καθημερινή βάση. Σας είπα ότι ενδεχομένως οι παρατηρητές και ορισμένοι συμμετέχοντες είχαν υποτιμήσει τα δεδομένα. Αυτό το είπα απαντώντας σε μια προγενέστερη ερώτηση. Και αυτό σημαίνει ε, ε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να ε, φτάσουμε σε μία δυναμική ε, πορεία, αναπτυξιακή πορεία. Αυτό το είπα και προηγουμένως και ισχύει για όλες τις χώρες και για τη Γερμανία. Η Γερμανία γνωρίζει μία ανάκαμψη η οποία ε, αφορά και την πρόοδο που έχει επιτελεστεί σε επίπεδα ανταγωνισμού. θα πρέπει να προωθήσουμε τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη γενικότερη οικονομική αναπτυξιακή πορεία. Αυτό αφορά μια γενική παρατήρηση για όλες τις χώρες χωρίς καμία εξαίρεση, διότι θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση αν είχαν γίνει αυτές οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η Σας ευχαριστώ που μας θυμήσατε ότι υπάρχουν και μερικά θετικά νέα για την οικονομία στον έξω κόσμο. Γιατί ακούμε τόσο <clears throat> αρνητικά και ανησυχητικά και τίνουμε να λησμονούμε και τα θετικά. Οι αγορές βέβαια εξακολουθούν και είναι πολύ ε, αναστατωμένες και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα λόγια που λέμε και τα μηνύματα που δίνουμε και ασφαλώς εγώ δεν θέλω να εξέλθω τη εντολή μου. Νομίζω μάλιστα ότι υπάρχει και υποχρέωση όχι μόνο των πολιτικών αλλά και των δημοσιογράφων να φροντίζουν να δίνουν και αυτοί πολύ καθαρά μηνύματα και ε, να μεταφράζουν ό,τι ακούν πολύ ε, ξεκάθαρα. Στην ε, στήλη λέξη των Financial Times, που είναι λίγο πολύ το κουτσομπολιό των χρηματαγορών σήμερα, λοιπόν στους Financial Times σχολιάζουν την συμφωνία που έγινε το Σαββατοκύριακο και λένε ότι μετά το 2013 ο μηχανισμός δεν θα, ε, σημαίνει, δεν θα επιφέρει haircuts, κουρέματα δηλαδή, εκτός εάν συμφωνήσουν οι υπουργοί ότι η κυβέρνηση, η θυγόμενη κυβέρνηση, ε, είναι αφαιρέγγια. Αυτά που βλέπω εγώ λοιπόν εδώ είναι ότι η δοκιμασία φερεγγιότητα θα γίνεται από την Κομισιόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όχι επομένω ομόφωνη απόφαση 27 ή έστω των 15 ε, ε, Υπουργών Οικονομικών. Περνούν λοιπόν το ε, τεστ φερεγγιότητα σε ανεξάρτητα χέρια. Ίσως αυτό είναι καλό για να σταματήσει αυτός ο πολιτικός καυγάς και Εάν αυτή είναι μια απόφαση που έλαβαν οι Υπουργοί Οικονομικών, πρέπει να δοθεί ξεκάθαρα ως μήνυμα προς τις αγορές. Όταν λοιπόν υπάρχει μια απόφαση, όταν λαμβάνεται μια απόφαση να μεταφέρεται πολύ καθαρά, να, να μεταφράζεται πολύ καθαρά και οι δημοσιογράφοι εφόσον έχουν ερωτήσεις, ας θέτουν τις ερωτήσεις πριν να τυπώσουν τα άρθρα τους. Τώρα έχω και ορισμένα άλλα ερωτήματα. <clears throat> Πρώτα, Είπατε ότι θα χαίρει ιδιαίτερου καθεστώτος ε, το δάνειο αυτό, δηλαδή μετά το 2013. Ή εφα, εφαρμόζεται ήδη και στην Ιρλανδία. Και για τις ρήτρες συλλογικών ε, δράσεων, για τι θα γίνει με τα ομόλογα, τα οποία θα έχουν ημερομηνίε μετά από το 2014 και βρίσκονται ήδη στα χέρια του κοινού, και τα ομόλογα που εκδίδονται από τώρα και μέχρι το 2013. Εγώ προτιμώ να μην κάνω εικασίε ε, σχετικά με το πώ θα ε, ρυθμιστεί το θέμα, αλλά προτιμώ να ακούσω την απάντησή σα. Ε, ευχαριστώ κύριε μου. <clears throat> Συμφωνώ με την πρώτη σας, ή τις πρώτες σας παρατηρήσεις. Δεν είναι ο καιρό κατάλληλο για συγκαταβατικότητα και χρειάζεται σαφήνεια, σαφήνεια, σαφήνεια. Είναι απόφαση των κυβερνήσεων. Έχουν την δήλωσή τους, όπως είπα, η δήλωση αυτή αποτελεί μια χρήσιμη διευκρίνηση. Υπάρχει λοιπόν τώρα αυτό το ε, κείμενο και πρέπει να προωθηθεί, να γίνει κείμενο επικοινωνίας όσο γίνεται καλύτερα. Όλες οι κυβερνήσεις επικοινωνούν. Μην ε, κατηγορούμε λοιπόν αδίκως ίσως τους δημοσιογράφους έχουμε ένα θέμα ότι ακούγονται πάρα πολλές φωνές. Αυτό είναι πρόβλημα, ναι. Και χρειάζεται απαραίτητο πειθαρχία στις φωνές αυτές. Σας ευχαριστώ και συμφωνώ μαζί σας. Ο Γκέι. Πρώτα σας ευχαριστώ για τις συμβουλές σας, κύριε Πρόεδρε, και δυστυχώς δεν ήσασταν παρόν στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα για να πείτε στον κόσμο να είναι ε, προσεκτικός με το τι λέει και δεν χρειαζόμαστε ταύρους ή αλλοπολία για τα θέματα, για τα θέματα της Ιρλανδίας. Κύριε Πρόεδρε, έχω να σας ρωτήσω το εξής. Μία πηγή στην Ιρλανδία ισχυρίζεται ότι πιέσατε την Ιρλανδική κυβέρνηση να δεχτεί τη δέσμη μέτρων και τώρα προχωρείτε στην άσκηση πίεσης στην Πορτογαλία. Εγώ δεν θα τολμούσα ποτέ να θέσω το θέμα αυτό, αλλά τα είπε αυτά ένας υπουργός και θα ήθελα, θα χαιρόμουν πολύ να άκουγα από εσά ότι δεν τους πιέσατε. Ναι, μεν ήσασταν επιτυχείς, ήταν επιτυχής η ε, προσπάθειά σας να τηρήσετε το βασικό σας στόχο, τη σταθερότητα των τιμών δηλαδή. Ο ίδιος μηχανισμός οδήγησε όσο σε πληθωρισμό των περιουσιακών στοιχείων, της ε, Ε, ιδιοκτησία, των ακινήτων δηλαδή. Δέχεστε κάποια από την ευθύνη για την κατάσταση αυτή, σε σχέση δηλαδή με, ένα πληθωρισμό των τιμών των ακινήτων και ποια είναι τα διδάγματα που αντλεί η ε, Κεντρική Τράπεζα για το μέλλον από την κατάσταση αυτή. Απάντηση του Πρόεδρου. Είναι σαφές ότι όταν μια χώρα ανήκει σε ένα χώρο ενιού νομίσματος διαστάσεων υπήρου και περισσότερο από 300 εκατομμύριων κατοίκων που είναι παραπάνω από τον αριθμό κατοίκων της, των Ηνωμένων Πολιτειών και όταν υπάρχει μια κεντρική τράπεζα με το καθήκον να εξασφαλίζει τη σταθερότητα τιμών σε αυτό το τεράστιο αριθμό οικονομιών στο σύνολό τους ακριβώς οι οικονομίες η οικονομία όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να γνωρίζουν ότι βρίσκονται, βρίσκονται ε, σε ένα πλαίσιο όπου βελτιστοποιείται η οικονομική σταθερότητα στο σύνολο των χωρών αυτών. Δεν μπορούμε να προσαρμόζουμε, ούτε μπορούσαμε να προσαρμόζουμε την ε, πολιτική μας οικονομική σταθερότητα, η νομισματική ένωσή μας, λαμβάνοντας μονάχα υπόψη τις ανάγκες της Γερμανίας, που ίσως θα μας ζητούσε πολύ χαμηλότερα επιτόκια κάποια στιγμή, που θα είχε όμως ως αποτέλεσμα πρόσθετες δυσχέρειες σε άλλες χώρες. Ούτε μπορούμε να προσαρμόσουμε την νομισματική μας πολιτική μονάχα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της Ιρλανδίας ή της Ισπανίας. Οφείλουμε να, να λάβουμε υπόψη, για παράδειγμα φέρνω σαν παράδειγμα το, το ισοδύναμό της από την Αλάσκα μέχρι τη Μασαχουσέτη για να εξασφαλίσουμε ε, νομισματική σταθερότητα για 320 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την ανάγκη αυτή και να κατανοήσουμε επίσης ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές, οι μακροπολιτικές συνολικά και στο βαθμό που εξαρτώνται από εθνικές αποφάσεις, οι πολιτικές εποπτείας, πρέπει όλες να είναι προσαρμοσμένες ώστε να λαμβάνουν αυτά υπόψη. Γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων ότι οφείλουν να σχεδιαστούν οι εθνικές πολιτικές με τρόπο ώστε πρόθεσμα ε, να βρίσκεστε γύρω στο 2% σε πληθωρισμό. Αυτό είναι το θέμα. Και με τον τρόπο αυτό ε, λειτουργήσαμε και εργαστήκαμε και δεν κάναμε και τίποτε άλλο. Αφού αν είχαμε ε, εργαστεί διαφορετικά θα πηγαίναμε από ένα μικρό μέρος του χώρου ευρώ σε ένα άλλο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το ίδιο όπως είπα για το ε, κόστος μονάδας εργασίας πρέπει να λάβουμε υπόψη που ακριβώς είναι το μέτρο για τα επόμενα 10 χρόνια, το benchmark. Δεν θα σχολιάσω τίποτε άλλο. Όλες οι κυβερνήσεις ε, προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποφύγουν σοβαρά σφάλματα, και να κινηθούν προς την σωστή κατεύθυνση διαρθωτικών δηλαδή μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής υγείας. Η Astrid Λούλινγκ. Κύριε Πρόεδρε, ένα θέμα που διαιρεί την Επιτροπή μας και θα συνεχίσει να διαιρεί ε, τις επόμενες εβδομάδες είναι το θέμα των ευρωομολόγων. Εγώ γνωρίζω το θεσμικό πρόβλημα που θέτει ο μηχανισμός αυτός, αλλά δεν θα συζητήσω αυτό. Θα ήθελα να μάθω μόνο από εσά για ποιο λόγο αυτά τα ευρωομόλογα δεν είναι κατάλληλα στο παρόν πλαίσιο, αφού οδηγούν σε μια ε, χαλάρωση ενώ χρειάζεται αυστηρότητα στην διαχείριση των δημοσίων οικονομικών των διαφόρων χωρών μελών. Και από την άλλη μεριά θα ήθελα να μάθω εάν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δεν ανταποκρίνεται ήδη σε ορισμένα κριτήρια των ευρωομολόγων. Έχουμε πράγματι ε, μια εγγύηση, έχουμε ένα ενιαίο ε, επιτόκιο. Πού βρίσκεται λοιπόν η θεμελιώδης διαφορά και τρεις ευχαριστίες ε, προς τον πρώτο Τρισέ. Πρώτον, διότι θυμήσατε πολύ καθαρά ότι το ευρώ διατήρησε την αξία του καλύτερα από τα άλλα νομίσματα. Ελπίζω ότι το μήνυμα αυτό ελήφθη. Ευχαριστώ επίσης που θυμήσατε τις μεγάλες ανησυχίες σας ήδη από το 2005 σχετικά με το Σύμφωνο της Σταθερότητας και για τον ε, ε, εντοπισμό των υπευθύνων αυτών των ε, βαρέων σφαλμάτων, την Ευρωμάδα δηλαδή, το Eurogroup. Ευχαριστώ επίσης για τα όσα κάνατε για θέματα σταθερότητας των τιμών, που αποτελεί την καλύτερη κοινωνική πολιτική για τα πιο αδύναμα στρώματα του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Σας ευχαριστώ για αυτές τις ευχαριστίες. Θα ήθελα απλώς να πω ότι αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα ύψης της σημασίας. Θα πρέπει οι κυβερνήσεις μας να δείξουν αποφασιστικότητα και να λάβουν υπόψη αυτή την αναγκαιότητα όχι μόνο να συμπεριφερθούν καλά, αλλά να υποπτεύσουν και τους άλλους. Γιατί δεν μπορεί κανείς να πει σε μια άλλη κυβέρνηση ότι δεν συμπεριφέρεται καλά, αλλά αυτό σημαίνει εποπτεία. Εποπτεία που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ως προς τα ευρωομόλογα ήδη απάντησα, εμείς δεν είχαμε ταχθεί υπέρ ποτέ. Τα ευρωμόλογα ε, αφορούν κοινέ εγγύησεις, ένα κοινό πλαίσιο εγγύησεων, διακρατικό και το Ευρωπαϊκό Τομείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, το EFSF, έλαβε ε, μία απόφαση για πρώτη φορά επί του θέματος. Αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως δεν έχουμε εκφέρει άποψη ούτε ως προς την κοινή έκδοση ευρωομολόγων με κοινό πλαίσιο εγγύησης ούτε για το 60% που αναφέρθηκε, γιατί αυτή ήταν μία από τις προτάσεις. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο πόλεμος των νομισμάτων δεν είναι επιθυμητός, εφόσον δεν είναι επιθυμητός. Δεν θα πρέπει να μιλήσουμε για διεθνή συνεργασία για να έχουμε ένα συνεκτικό νομισματικό σύστημα. Τρεις ερωτήσεις. Σε σχέση με τους G20 χρειάζεται μία μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος. Πώς θα συνεισφέρει η ΕΚΤ. Ως προς τις αναδιόμενες χώρες θα πρέπει να έχουν μετατρέψιμα νομίσματα και αυτό δεν πρέπει να γίνει βαθμιαία. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει νοθρότητα. Συμφωνείτε με αυτό το κριτήριο της μετατρεψιμότητας και σε σχέση με τη σταθερότητα τιμών μας έναντι των ΗΠΑ, πιστεύετε ότι η νομισματική μας πολιτική είναι συμβατή με τα συμβατικά και μη συμβατικά μέτρα που έχει εγκρίνει η ΕΚΤ και πώς συσχετίζεται αυτό το θέμα με τη ΦΕΔ. Thank you very much Σας ευχαριστώ. Ως προς το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα, αυτό που μετράει είναι η περίπλοκη φύση των ε, διακυβευμάτων, εγώ είδα δύο διαφορετικά ζητήματα. Τα κειμενόμενα νομίσματα μέσα στα πλαίσια ενός μονίμου καθεστώτος από τότε που έληξε το σύστημα Bretton Woods, δηλαδή από τη δεκαετία του 70 και βεβαίως έχουμε να κάνουμε και μετανομίσματα των αναδιωμένων χωρών. Αυτό είναι το δεύτερο σας ερώτημα και θα ήθελα να πω, να απαντήσω καταφατικά. Οι εν λόγω χώρες έλαβαν μία απόφαση. Ίσως πρόκειται για μία βαθμία και εντάξει διαδικασία, έτσι ώστε τα νομίσματα αυτά να ενταχθούν ε, βαθμία σε, μια, ε, γενικότερη, σε ένα γενικότερο ευέλικτο πλαίσιο. Οι G20 αναφέρθηκαν σε αυτό το σημείο και αυτό ε, αντικατοπτρίζει μία παγκόσμια διαδικασία συνένεσης. Βέβαια είναι ευκολότερο το να λεχθεί παρά να γίνει κάτι τέτοιο. Ως προς το τρίτο σας θέμα, θα πρέπει να πω ότι μαζί με το ΦΕΔ έχουμε αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης και φιλίας και χωρίς αυτή τη συνεργασία με την ΦΕΔ δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την δυνατότητα να αντισταθούμε στην κρίση όπως κάναμε το 2008 και 2009. και με τη δυνατότητα που ε, δόθη από την ΦΕΔ παροχής ρευστότητας δολαρίων μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας Ανταλλαγών, Swap Agreement. Είναι κάτι που θεωρώ ως ένα πολύ βασικό στοιχείο σε διεθνές επίπεδο, ότι υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μεγάλων κρατικών τραπεζών. Αυτό αφορά και την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας, της Ιαπωνίας, των ΙΠΑ Και αυτό αφορά και τις αναδυόμενες χώρες θα κάνω κάτι που δεν κάνω συχνά. Θα πω κάτι στο τέλος της συνεδρίασής μας. Είπατε κάτι επανάληψη. Ότι δεν επιθυμείτε να <clears throat> ανατραπεί ένας επιτυχής μηχανισμός σταθερότητας και αυτό βεβαίως το επιθυμούν και πολλά μέλη της παρούσας Επιτροπής και ίσως να μην θέλετε να σχολιάσετε τα όσα θα πω εγώ τώρα, αλλά εκπλήσωμαι στο πλαίσιο των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Ε, ευνηδιάζομαι από την ισορροπία των πόρων που λαμβάνονται από τον προϋπολογισμό και τον δημοσιονομικό μηχανισμό Και μου φαίνεται ότι από τις αγορές παίρνουμε πολύ λίγα χρήματα ε, για το ταμείο αυτό, που ίσως να είναι εσφαλμένο προηγούμενο. Με ανησυχεί όταν βλέπω και τα επιτόκια που κυκλοφορούν και που ίσως είναι λιγότερο ευνοϊκά από του ε, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. <clears throat> Αν και κατανοώ βέβαια την ανάγκη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, δεν θεωρώ ότι είναι σόφρον αυτό. Στις μελλοντικέ συναντήσεις ελπίζω ότι αυτές οι ανησυχίες με κάποιο τρόπο θα αντιμετωπιστούν. Θα συζητηθούν δηλαδή. Διότι αλλιώ φοβούμαι ότι θα υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι θα υψώσουν τις, φωνές, τις φωνές ανησυχίας τους, κυρίως σε ό,τι αφορά την διαδικασία με την οποία ελήφθησαν οι αποφάσεις αυτές, και που ίσως να μην είναι απόλυτα διαφανής η τρόπη αυτοί. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε σε ορισμένες από αυτές τις σκέψεις μου και βέβαια την επόμενη εβδομάδα θα διευκρινιστούν τα του ε, μηχανισμού επιτοκίων. Πρόεδρος Τρισέ, ευχαριστώ για τις παρατήρησεις που κάνατε και το ε, υπονοούμενο ερώτημά σας. Κάθε αρχή, κάθε θεσμός θα πρέπει να έρθει στο ύψος των ευθυνών του. Το είπαμε από την αρχή. Εμείς προσπαθούμε να αρθούμε στο ύψο των ευθυνών μας. Εξηγήσαμε και στο Κοινοβούλιο τι ακριβώ πράττουμε και τι είδου προσπάθειες νομίζουμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε. Και αυτό ισχύει για όλε τις αρχές και όλους τους θεσμού, όλα τα θεσμικά όργανα. Η διαρκή μα συμβουλή είναι αυτή τη στιγμή αποφασίσατε να δημιουργήσετε ένα μηχανισμό, ένα ταμείο το EFSF εν προκειμένου, προσπαθήστε να είστε όσο, δυνα, όσο το δυνατόν πιο εύκαμπτοι και να προσφέρετε τη μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια. Αυτό μου φαίνεται κοινή λογική. Αλλά βέβαια, σέβομαι το γεγονός ότι και οι κυβερνήσεις και εθνικά κοινοβούλια έχουν τους δικούς τους κανόνες, έχουν τις δικές τους οπτικές και όπω είπα πρέπει να είμαστε ε, ε, ταπεινόφρονες ε, μπροστά στους νόμους αυτού τη δημοκρατία μα. Εάν όμω όπω είπα, αποφασίσετε τελικώς να δώσετε τη βοήθεια αυτή, να είστε εύκαμπτοι και να δώσετε τη μέγιστη δυνατή βοήθεια που ε, υποβάλλουν οι περιστάσεις, υπογορεύουν οι περιστάσει. Εάν το αποφασίσετε εν τέλει. Γενικότερα θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. όπω είπα, δεν πρέπει να είμαστε σκεταβατικοί. Χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο προσανατολισμό. Και πιο γενικά και μιλώ μάλιστα και για λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και για το Κοινοβούλιο το ίδιο. Πρέπει να ενισχύσουμε την ε, εξουσία εντό εισαγωγικών των ε, δημοσίων αρχών. Γιατί στην βάση αυτής μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις απαιτήσει αυτές που θα είναι πολύ απαιτητικές οι περιστάσεις και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τα σχόλια σας αυτά, λέει Πρόεδρος. Εδώ <clears throat> λίγη η ε, συνάντηση αυτή του νομισματικού διαλόγου και θα ξεκουραστείτε λίγο με τον επόμενο Μάρτιο, αν και νομίζω ότι θα συναντηθούμε ξανά πολύ συντομότερα. Είναι ένα πολύ καλό